Bene. Buongiorno a tutti. Καλημέρα σας. Μπορούμε να ξαναρχίσουμε τις εργασίες της Επιτροπής μας. Αρχίζουμε με το πρώτο θέμα της ημερήσιας ε, διάταξης που αφορά την έγκρισή της. Εάν δεν υπάρχουν ε, αιτήματα από τους συναδέλφους θεωρούμε ότι εγκρίνεται η μερίσια διάταξη χωρίς αλλαγές. Ως προς το θέμα υπαριθμών 2 έχω μία ανακοίνωση σε σχέση με, την, με τις αλλαγές σε ορισμένα σημεία ως προς τη σειρά δηλαδή συζήτησης ορισμένων θεμάτων. Το 4 της συναδέλφου Νίμπλερ που αφορά την διαστημική βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αλλάξει με το 9 της συναδέλφου Φόρντ. Επίσης υπάρχει ένα άλλο ζήτημα για το οποίο θα ήθελα να σας πληροφορήσω που αφορά τις τροπολογίες έκθεσης Βιντάλ Κουάδρας η Επιτροπή ΕΜΒΗ δεν δέχτηκε τις τροπολογίες της Ήτρε ε, σε σχέση με την έκθεση Βιντάλ Κουάδρας. Ήρθαμε σε επαφή με τους συντονιστές γραπτός, γιατί δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα και συμφωνήσαμε να υποβάλουμε τις τροπολογίες στην Ολομέλεια δυνάμει του άρθρου 50. Η πλειοψηφία των συντονιστών τάχθηκε υπέρ της πρότασης αυτής και συνεπώς οι τροπολογίες που δεν εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Περιβάλλοντος θα υποβληθούν στην Ολομέλεια, εξ ονόματος της Επιτροπής μας. Αυτή είναι η πληροφόρηση, η πληροφορία που ήθελα να σας δώσω. Η κυρία Στότερ. Ευχαριστώ. Θέτω υπόψη σας ότι η ομάδα των πράσινων είναι αντίθετη με την κατάθεση τροπολογιών για την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Δεν συμφωνούμε με την πρόταση αυτή. Ευχαριστούμε την ε, συνάδελφο, θα το λάβουμε υπόψη. Είπα ότι αυτό ε, έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία και έτσι θα πρέπει να το δεχτούμε. Βιντάλ Κουάδρα, σε σχέση με αυτό το ζήτημα που θίξατε, θα πρέπει να πω ότι την τελευταία εβδομάδα έγιναν πολλές συναντήσεις μεταξύ μου και της κυρίας Λεπάζ, της εισηγήτριας και καταβάλαμε μεγάλες προσπάθειες για να συμφιλιώσουμε τις θέσεις και των δύο επιτροπών προσπαθώντας να φτάσουμε σε μία ε, ισορροπημένη άποψη έτσι ώστε να συγκλίνουν οι θέσεις των δύο επιτροπών. Δυστυχώς, δυστυχώς όμως οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Αφορούν ε, σημεία μείζωνος σημασίας, γι' αυτό δεν μπορούν να επιληθούν εύκολα. Καταβάλαμε μεγάλες προσπάθειες η κυρία Λεπάζ και εγώ, αλλά δεν επιτύχαμε. Οι 45 τροπολογίες εγκρίθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία από αυτή την Επιτροπή και η Επιτροπή Περιβάλλοντος δέχτηκε μόνο δύο από τις 45. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να υποβάλουμε τις δικές μας τροπολογίες της Επιτροπής Ήτρε στην Ολομέλεια, αλλά θέλω να τονίσω ότι καταβάλαμε μια ειλικρινή και σοβαρή προσπάθεια μέχρι τέλους. Δυστυχώς όμως δεν στάθηκε δυνατό να φτάσουμε σε συμφωνία. Ωραία, ευχαριστώ τον συνάδελφο Βιντάλ Κουάδρας. Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης που άλλαξε με το 4 και θα ήθελα να δώσω το λόγο στη συνάδελφο Φόρτ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και ελπίζω όλοι να περάσετε καλές διακοπές και ευχαριστώ την κυρία Νίμπλερ που δέχτηκε την αντιστροφή των σημείων μα στην ημερήσια διάταξη για να προλάβω να πάω και σε άλλη επιτροπή που έχω έκθεση. Και περιμένω με ανυπομονησία τις απόψεις των σχεδόν εισηγητών για την γνωμοδότησή μου, που μάλιστα συνέταξε λίγο πριν τι θερινέ διακοπέ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή της Επιτροπής Περιβάλλοντος, τον κύριο Κρίς Ντέιβις, που διοργάνωσε μια σειρά σεμιναρίων και δυνατότητες επαφή και με τη βιομηχανία και με ακαδημαϊκούς ώστε να ενημερωθούμε και να διαμορφώσουμε τεκμηριωμένη άποψη πριν την κατάρτιση της έκθεση. Και θα έχουμε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εμείς βέβαια, επικεντρωνόμαστε σε θέματα ενέργειας κυρίως. Κάνοντας και τη δική μου έρευνα για την γνωμοδότηση, εντόπισα τρία ουσιώδη σημεία που μου τα επισήμαναν ως νευραλγικά και οι εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτό. Πρώτον, αν θέλουμε σοβαρά ένα, μια ασφαλή πηγή ενέργειας και αξιόπιστη και να μειώσουμε τον αριθμό των καυσερίων που διοχετεύουμε στην ατμόσφαιρα, ο, ο μόνος τρόπος και η μόνη τεχνολογία μεγάλης κλίμακας που έχουμε διαθέσιμη και που μπορεί να απομακρύνει το, να ξεπίσει το ανάθρακα από την καύση των ορυκτών καυσίμων και να το χρησιμοποιήσει για παραγωγή ενέργειας είναι η μέθοδος δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα. Εξετάσαμε διάφορες άλλες βιομηχανικές μεθόδους που δεν απέβησαν βιώσιμες ή φιλοπεριβαλλοντικές. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτό το σύστημα, το CCS, της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, γιατί αλλιώ θα παρακολουθήσουμε τις προσπάθειές μας και εθνικά και παγκόσμια προκειμένου να ε, αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Και η Ευρώπη δυστυχώς υστερεί σε σχέση με άλλες περιοχές του πλανήτη, γιατί ακούσαμε για αντίστοιχα προγράμματα στον Καναδά, ε, στην Κίνα και μάλιστα κάποιοι συνάδελφοι επισκέφθηκαν ε, τη χώρα αυτή. Φαίνεται ότι η Ευρώπη υστερεί σε θέματα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα δεν έχουμε αξιοποιήσει πλήρως ε, το δυναμικό μας. Και υστερούμε ε, από τους υπόλοιπους στον κόσμο. Μία τέτοια όμως υστέρηση διακυβεύει την βιομηχανική μας ανταγωνιστικότητα. Επίσης, ε, όπως πολλοί μου επισήμαναν, ένας από τους λόγους που ίσως δεν επενδύουμε ή δεν επιδιώκουμε να προσελκύσουμε επενδύσει στη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και σε άλλε τεχνολογίε με χαμηλή χρήση άνθρακα είναι επειδή ακριβώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει του δικού τη ε, ειδικού στόχου για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. και θέλει να απορροφήσει επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υποβαθμίζοντας τις επενδύσεις σε άλλες τεχνολογίες με χαμηλή χρήση άνθρακα. Αυτό που επιθυμίζω στην γνωμοδότησή μου είναι να θυμηθούμε τα πλεονεκτήματα μιας προσέγγισης ε, τεχνολογικά ουδέτερης ό,τι αφορά την ε, παραγωγή ενέργειας με χαμηλή χρυσή άνθρακα εν ώψη του ορίζοντα 2030. Είναι σημαντικό αυτό όταν θα θεσπίσουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους μας, να είμαστε τεχνολογικά ουδέτεροι και να μην μεροληπτούμε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε μπορούμε να επενδύσουμε και σε άλλες τεχνολογίες χαμηλής χρήσης άνθρακας, όπως είναι η δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα. Δεν υποβαθμίζω τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά θα, πρέπει αυτές να μονοπολίσουν το ενδιαφέρον. Αυτά και περιμένω τις απόψεις και των υπόλοιπων σχεδόν εισηγητών. Ευχαριστώ. Bene, ε, Ο κύριος Ντέιβις έχει το λόγο που είναι εισηγητής από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Όπως είπατε και εσείς είμαι εισηγητής περιβάλλοντος και έρχομαι εδώ σε κάποια κατάσταση αμηχανίας διότι άκουσα ότι ε, μόλις ότι η Επιτροπή μου δέχτηκε μόνο δύο από τις 45 δικές σας τροπολογίες. Πάντως δεν ευθύνομαι εγώ. Αισθάνομαι κάπως τόσο δημοφιλής όσο ένας που αποφεύγει το ποτό και πηγαίνει τώρα να επισκεφθεί ε, ένα ποτοπίο θα πρέπει να συνεργαστούν οι επιτροπές. Προ πενταετίας είχαμε μεγάλες ελπίδες για την ανάπτυξη του CCS. Είχε πει το Συμβούλιο ότι μέχρι το 2015 θα θέλει 12 μεγάλα έργα και το Κοινοβούλιο μάλιστα είχε προβλέψει και χρηματοδοτικό μηχανισμό για να συνδράμει τις χώρες να προωθήσουν τα συστήματα αυτά σύλληψης και αποθήκευσης του άνθρακα. 2013 σήμερα όμως δεν έχουμε τίποτα να δείξουμε προχωρήσαν 13 έργα με τη χρηματοδότηση αυτή, κανένα όμως δεν έχει μπει στην πρώτη φάση λειτουργίας. Ορισμένα από αυτά αποσύρθηκαν μάλιστα, για διαφόρους λόγους και κυρίως διότι ενώ δίνουμε χρήματα των φορολογουμένων και τους δίνουμε επιδοτήσεις για ανανεώσιμες ενέργειες, το CCS εξαρτάται αποκλειστικά από την τιμή του άνθρακα για να προχωρήσει και ξέρουμε πού έχει φτάσει η τιμή αυτή. Αυτό που βλέπω σήμερα είναι ότι κινδυνεύουμε να μην προωθήσουμε το CCS, που είναι όμως η μοναδική τεχνολογία η οποία μπορεί να αφαιρέσει το, ναι, το διοξείδιο του άνθρακα που εκλείουν διάφορες βιομηχανίες, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιμα χωρίς να υπάρχει η συνέπεια της θέρμανσης του πλανήτη. Και βεβαίως τα ορυκτά καύσιμα σε ολόκληρο το πλανήτη συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται και να καίονται. Και όλες οι μελέτες δείχνουν ότι το CCS θα είναι λιγότερο δαπανηρό από, ακόμα και στα πρώτα του χρόνια λειτουργίας, από την αιωλική ή την ηλιακή ενέργεια. Και υπάρχει μεγάλη ε, δυνατότητα αποθήκευσης για πολλά χρόνια για όλο το διοξίδιο άνθρακος που εκκλείεται στην Ευρώπη. Είχαμε, ήμασταν στην πρωτοπορία προ λίγων ετών. Τώρα καθυστερούμε, μένουμε όλο και πιο πίσω απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, τον Καναδά και ούτω καθεξής. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει. Πρώτα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι εδώ οι βασικοί παίκτες είναι οι χώρες μέλη. Αν θέλουν οι χώρες μέλη να βάλουν στο, στο χαρτοφυλάκια τους το CCS, τότε να το κάνουν. Μπορούν να βρουν τα χρήματα και θα πρέπει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο. Αν μια χώρα μέλος δεν θέλει να δεχθεί, να υιοθετήσει το CCS, Κανένας δεν πρόκειται ωστόσο να επενδύσει σε μια χώρα όπου δεν θα έχει με το πλευρό του την κυβέρνηση. Δεν θα ενδιαφέρεται δηλαδή η κυβέρνηση να προωθήσει το CCS. Στην Ευρώπη διαρωτώ αν κάποιες κυβερνήσεις το έχουν κάνει σκεφτεί το θέμα. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να υπάρξει νομική δέσμευση για τις χώρες μέλη να καταθέσουν ενδεικτικούς οδικούς χάρτες για το πώς θα εκπληρώσουν τους στόχους τους για το CCS, για την αποθήκευση του άνθρακα. Οι ΔΕΜΗ πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά, ε, οι στόχοι αυτοί. Τι μπορούμε να κάνουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει πρώτα να αρχίσουν να λειτουργούν κάποια έργα, κάποια πιλωτικά έργα. Δεν φτάνουν όμως αυτά. Χρειαζόμαστε ολόκληρη την αντισίδα σύλληψης και δέσμευση δηλαδή και αποθήκευση του άνθρακα και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να προβούν τουλάχιστον σε μια διακήρυξη ρεαλιστική 1,5 γιγαβάτ παραγωγής ρεύματος που να έχουν τα εργοστάσια που παράγουν το ποσό αυτό της ενέργειας να έχουν και συστήματα δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα μέχρι το 2020. Και βεβαίως, όπως λέει και η Βίκη Φόρτ στην έκθεσή της, θα συνδράμει σημαντικά στην προσπάθεια αυτή αν αυτά οι εμβληματικές ενέργειες μπορούν να ενταχθούν μέσα στους στόχους των ανανεώσιμων. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Βεβαίως το CCS δεν είναι ανανεώσιμη ενέργεια, όμως θα ενθαρρύνει τις χώρες μέλη να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να δώσουν χρήματα. Και όσοι ασχολούνται σοβαρά με την καταπολέμηση της θέρμανσης του κλίματος θα συμφωνήσουν. Τέλος, για το core funding, για την χρηματοδότηση. Πρώτα, για τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση. Πιστεύω ότι ο ορίζοντας του 2020 δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε ένα ταμείο για την βιομηχανική καινοτομία. Κάτι που να μπορεί να υποστηρίξει καινοτόμες ανανεώσιμε ενέργειες, όπως έγινε και με το EAR ε 300. Διακομματικά εμείς υπερψηφίσαμε στο Κοινοβούλιο, αλλά κάπου ανακατεύτηκε με το λεγόμενο backloading. Χρειάζεται να επανέλθουμε στην προσπάθεια αυτή. Εν τέλει, μακροπρόθεσμα, κυρία Πρόεδρε, νομίζω πρέπει να κινηθούμε και προς την κατεύθυνση έκδοσης πιστοποιητικών CCS από το 2020 και μετά. Διότι ο άνθρακας και, και τα άλλα οι βιομηχανίες το χρησιμοποιούν αυτά, δηλαδή βγάζουν λεφτά διοχετεύοντας στην αγορά καύσιμα τα οποία εκλείουν άνθρακα, α, ε, διοξείδιο του άνθρακα δηλαδή. Πρέπει λοιπόν να βάλουν και αυτοί το χέρι στην τσέπη για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Το Συμβούλιο ωστόσο δεν λέει τίποτα, δεν λέει καθόλου πώς θα προχωρήσουμε. Ζητώ λοιπόν από το Κοινοβούλιο και από την παρούσα Επιτροπή να συνδυάσει τις προσπάθειές της με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, να δούμε πώς μπορούμε να επαναφέρουμε το θέμα στην ημερήσια διάταξη και να το συνδυάσουμε με νέες ιδέες για την πρόθεσή του. Θα πρέπει να ανακτήσουμε λίγο το χρόνο μας, το χαμένο χρόνο, γιατί ε, χάσαμε λίγο χρόνο. Ο κύριος ε, Μαρτσιβιέβιτς για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια στην Ευρώπη για τη μείωση του διοξιδίου του άθρακα προκειμένου να συμβάλλουμε στην παγκόσμια προσπάθεια καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. Οι αναπτυγμένε χώρε όμω και οι αναπτυσσόμενε χρειάζονται ενέργεια για να αναπτύξουν τη βιομηχανία του. Οπότε η κατανάλωση ενέργεια θα αυξηθεί στο μέλλον. Και φαντάζομαι πολλέ αναπτυσσόμενε χώρε ε, θα χρησιμοποιήσουν ε, ορυκτά καύσιμα. Άλλωστε ε, είναι σημαντική πηγή άνθρακα, Βέβαια δεν θα πρέπει η χρήση του άνθρακα να υποβαθμίσει του στόχου μα για τη μείωση των καυσαερίων σε ό,τι αφορά την δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Έχουμε, είχαμε για πολλά χρόνια ε, μια άνθηση αυτής της ε, προσπάθειας ε, και, κάποιες, και κάποια σημαντικά προγράμματα, αλλά φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε ευθύνουσα πια πορεία σε ό,τι αφορά τη μέθοδο αυτή. Θα πρέπει να δοθούν κάποιες εγγυήσεις από τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Γιατί διάφορα μοντέλα και προγράμματα που έγιναν ε, για, τον, την τεχνολογία αυτή ήταν περισσότερο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν έχει φτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η τεχνολογία σε αρκετό όριμο στάδιο ώστε να μπορούμε αξιόπιστα να προβλέψουμε ε, την ε, γενικευμένη εφαρμογή της και μάλιστα σε το χρόνο. Για να έχουμε εμπορική δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστούμε τεράστιες επενδύσεις, ε, μεγάλο κόστος και δεν υπάρχουν και εγγυήσεις για την αποτελεσματικότητα και την οικονομική αποδοτικότητα ενός τέτοιου προγράμματος. Θα πρέπει να αναπτύξουμε τις τεχνολογίες μας, αλλά δυστυχώς δεν δόθηκαν αρκετά ενάυσματα όπως το NER 300 για να αναπτυχθεί αυτή η τεχνολογία. Και μάλιστα ε, χρειάζεται περισσότερο να έχουμε μικρής κλίμακας και πολύ περισσότερα προγράμματα ε, αποθήκευσης και δέσμευσης του άνθρακα παρά λίγα και πολύ μεγάλα, μεγάλης κλίμακας προγράμματα. Τώρα, αν έχουμε θετική έκβαση τέτοιων μικρών προγραμμάτων, μπορούμε να περάσουμε σε μια πιο εμπορική εκμετάλλευση της τεχνολογίας αυτής. Ε, στο μέλλον θα πρέπει να δούμε αν πραγματικά είναι ε, εμπορικά αποδοτικό αυτό το σύστημα και φυσικά χρειαζόμαστε και ενημερωτική εκστρατεία ε, για την, για την κοινή γνώμη, γιατί μερικές φορές το ευρύ κοινό αγνοεί την, τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας και επίσης δεν είναι και γνωστές μερικές μέθοδοι γεωλογικής αποθήκευσης του άνθρακα. Χρειάζεται λοιπόν καλύτερη ενημέρωση. Σίγουρα όλοι χρειαζόμαστε πιο φθηνή ενέργεια και ε, αυτή τη στιγμή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς άνθρακα είναι το 30% της Ευρώπης. Έχουμε εκτεταμένη χρήση, θα πρέπει να εφαρμόσουμε όμως πιο αποτελεσματικές μεθόδους ε, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και παραγωγής θερμότητας. Φυσικά θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε τις εγκαταστάσεις ε, με χρήση ορυκτών καυσίμων προκειμένου να έχουμε λιγότερα καυσαέρια ε, για το περιβάλλον και να έχουμε πιο φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους όπως είναι αυτή τη συνδέσμευση και ε, αποθήκευση του άνθρακα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς έχουμε πολύ ακριβή ενέργεια. Θα πρέπει να μειώσουμε την τιμή της και η χαμηλή τιμή ενέργειας θα πρέπει να είναι βασική προϋπόθεση για τη χρήση νέων τεχνολογιών. Ευχαριστώ, η κυρία Χέρτσοκ. Συγγνώμη, Πρόεδρε, που άργησα. Θεώρησα ότι θα συζητηθεί αργότερα το θέμα. Ως σκιώδης από ότι τους σοσιαλιστές, σοσιαλιστές θα ήθελα να σας πω ποια είναι η άποψή μας και να υποβάλω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η θέση των σοσιαλιστών σε σχέση με την πράσινη τεχνολογία ε, ορίζεται στο έγγραφο ενεργειακής πολιτικής και που θα πρέπει να διαβάσω. Η δέσμευση και αποθήκηση του άνθρακα θα μπορούσε να ήταν χρήσιμη όταν χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιμα και λάβουμε υπόψη και τις βιομηχανικές ε, εκπομπές γενικότερα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι χρειάζονται, χρειάζονται μελέτες, ε, μελέτες αντικτύπων. Αυτή είναι η ευρύτερη θέση των σοσιαλιστών για την δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα, ιδιαίτερα όσον αφορά την χρήση βιομηχανικών μονάδων. Συμφωνήσαμε με την τεχνολογία CCS μετά από την προϋπάρχουσα ε, κρίση και θα πρέπει η νομοθεσία και ιδιαίτερα η οδηγία για τη δέσμευση και αποθήκευση, να λάβουμε υπόψη ότι επιβραδύνθηκε η διαδικασία γενικότερα με βάση τη νομοθεσία. Θεωρούμε λοιπόν ότι χρειάζεται μία έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Η ερώτησή μου προς την Επιτροπή είναι η εξής. Στο σχέδιο ανάκτησης Έχουμε θέσει ένα δις ευρώ για τα προγράμματα επίδειξης και θα ήθελα να ρωτήσω τι συνέβη με αυτό το ένα δις, πώς δαπανήθηκε και αν όχι γιατί. Και αν δεν δαπανήθηκαν τα χρήματα, πού βρίσκονται, πώς ε, και τι μπορούμε να κάνουμε για να δαπανηθούν αυτά τα χρήματα τον υπολοιπόμενο χρόνο γιατί η αύξηση των ορυκτών καυσίμων είναι μεγαλύτερη. Ε, ζητάμε καθαρές τεχνολογίες αποθηκευσής και δέσμευσης γενικότερα και από πλευρά σοσιαλιστών θεωρούμε ότι η χρηματοδότηση είναι σοβαρό θέμα. Δεν θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει χρηματοδότηση από τον ορίζοντα 2020, αλλά από το σύστημα EPS. Θα πρέπει όμως να βρούμε τη σωστή χρηματοδότηση έτσι ώστε οι χώρες που εμπλέκονται άμεσα της δέσμευσης και αποθήκευσης να τεθούν χωριστά σε σχέση με εκείνες που δεν εμπλέκονται στο σχέδιο CCS. Θέλουμε να υπάρξει μια ευελιξία και να δούμε πώς το σχέδιο ε, ανταλλαγής εκπομπών μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα ή έμεσα. Τέλος, εάν πρέπει, αν φτάσουμε στον ποσοστιαίο στόχο που έχουμε ορίσει, θα πρέπει να προωθήσουμε το θέμα άμεσα. Εάν δεν μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο θα πρέπει να πούμε και στους Ευρωπαίους πολίτες ότι δεν καταφέρνουμε ε, να αντιμετωπίσουμε το θέμα της, ε, της αντιμετώπισης της θερμοκρασίας και της μείωσης κατά δύο βαθμούς. Πρώτη, νομίζω ότι το θέμα της ε, δέσμευσης και αποθήκευσης εμπλέκεται στα δύο τρίτα εκπομπών. Άρα δεν έχει και τόσο ε, μεγάλο νόημα όπως το αντιμετωπίζουμε εδώ, διότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε θέματα καύσης ή αποφυγής καύσης. για να φτάσουμε σε μια πραγματική και, θετική, και θετικό διαχωρισμό του άνθρακα θα πρέπει να ξέρουμε πού υπάρχει διάχυση, στη γη μέσα στα πλαίσια της εξοικονόμησης υδάτινων πόρων και της χρησιμοποίησης των γεών. Ευχαριστούμε. Μπρετζίνα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγητριά μας για την πολύ καλή της γνωμοδότηση, στην οποία μάλιστα καλύπτει όλες τις πτυχές αυτής της τεχνολογίας που μας ενδιαφέρει και τη υστέρησης ε, που παρατηρούμε στην Ευρώπη ως προς εξελίξη την τεχνολογία αυτή. Παρακολούθησα στην Κίνα τις προσπάθειες που γίνονται με επίσκεψη που έκανα εκεί και είδα ότι όλα τα τεχνολογικά στοιχεία αυτών των εγκαταστάσεων ε, είναι πολύ πιο προηγμένα. Έτσι γίνεται πλήρης αξιοποίηση των και παραγωγή 200 ΜΒ. Η επόμενη γενιά των τεχνολογιών αυτών ε, θα αναγκαστεί να χρησιμοποιεί κινέζικα προϊόντα. Ενώ στην ε, Ευρώπη χάνουμε όλο και περισσότερο έδαφος και βρισκόμαστε όλο και, όλο και πιο πίσω. Σε ό,τι αφορά την δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα, πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε γιατί ποσότητα ενέργειας μιλάμε. Η Κινέζοι παραγωγοί και κατασκευαστές ε, μας μιλούν για πολύ διαφορετικά αριθμητικά στοιχεία από αυτά που εξετάζουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις νέε τεχνολογίες γιατί είναι σημαντικές όχι μόνο από εμπορική άποψη, αλλά και λόγω της ε, μεταβαλλόμενης κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνάδελφο Βίκη Φόρτ για την πολύ καλή της γνωμοδότηση και να πω ότι εμείς δεν είμαστε κατά του CCS, της δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα. Δεν υπάρχει διχασμός μεταξύ μας. Είμαστε υπέρ των τεχνολογικών καινοτομιών. Αλλά δυστυχώς βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση και βαδίζουμε σημειωτών ε, εδώ και πολλά χρόνια. Δεν έχουμε σημειώσει καμία πρόοδο. Χρειάζεται, χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις και το κόστος αυτό θα πρέπει να το αναλάβουν οι κυβερνήσεις. Αλλά φαίνεται ότι και η κοινή γνώμη είναι κατά αυτού του συστήματος, γιατί δεν φαίνεται να είναι αποδοτική αυτή η τεχνολογία και δεν φαίνεται να υπάρχουν και δυνατότητες ανάπτυξής της γιατί όπου και αν δοκιμάστηκε η τεχνολογία αυτή οπουδήποτε και αν έγιναν απόπειρε εφαρμογής της ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε ανησυχία στο ευρύ κοινό τι θα γίνει με αυτή την ορολογιακή βόμβα ε, φοβάται ο λαός και ε, ο κόσμος και είναι δύσκολο να εξηγήσουμε στον κόσμο τι θα γίνει με, αυτό το τον αποθηκευμένο άνθρακα. Ο κόσμος δεν γνωρίζει την κατάσταση και φοβάται πολύ. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ε, ενημερώσουμε καλά τον κόσμο και να είμαστε πολύ προσεκτικοί ιδιαίτερα γιατί στην Ευρώπη έχουμε πολύ πυκνοκατοικημένες περιοχές. Επίσης, θα ήθελα να αναβερθώ στο, στη δεύτερη ε, αιτιολογική σκέψη. Στο Β λέει η συγγετριά μας ότι το CCS αφορά μόνο την παραγωγή ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας. Διαφωνώ. Δεν αφορά μόνο την παραγωγή ενέργειας το CCS, αλλά και τη χημική βιομηχανία, ε, τα λοιπάσματα, τη βαριά βιομηχανία. Πρόκειται για τεχνολογία δηλαδή που μπορεί να είναι αποτελεσματική και λειτουργική για πάρα πολλά χρόνια, άσχετα με τις αλλαγές στην ενέργεια και στο κλίμα. Αρκεί φυσικά να, περάσουμε, να ξεπεράσουμε το σημαντικότερο εμπόδιο στη χρήση αυτής της τεχνολογίας που είναι αυτή τη στιγμή κοινή γνώμη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει κανείς να εξετάζει στην παραγωγή ενέργειας ολόκληρη την αλυσίδα από εκεί όπου εξορίσεται το καύσιμο στην περίπτωση αυτή μέχρι με τον πιο τρόπο γίνεται η καλύτερη εκμετάλλευσή του. Και το διοξίδιο του ανθρακός είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη βιομηχανική διαδικασία παραγωγής διαφόρων προϊόντων. Άρα δεν είναι μόνο η αποθήκευση που πρέπει να μας απασχολεί στη συζήτηση αυτή ενδιαφέρει για παράδειγμα υπάρχει και ο Ούγκρος νομπελίστας που διαπίστωσε ότι διοξείδιο του άνθρακα και νερό σε συνδυασμό αποδίδουν μεθανόλη. Μπορεί λοιπόν να, μπορούν να βελτιωθούν αυτές οι διαδικασίες που επιτρέπουν την βελτίωση της εκμετάλλευσης της, ε, του προϊόντος και να περιληφθούν στις διαδικασίες αυτές οι διάφορες, ε, ε μάλλον στην παραγωγή και στην εκμετάλλευση του αέριου. Ο κύριος Βιδάν Προέδρας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφυσβήτητα η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην πορεία προκειμένου να έχει ένα πιο ασφαλές ε, σύστημα παραγωγής ενέργειας, αξιόπιστο και ε, φιλοπεριβαλλοντικό. Αξιέπαινοι αυτή η στόχοι, καταπληκτική, αλλά για την υλοποίησή τους χρειαζόμαστε διάφορες τεχνολογίες και ε, διαφορετικές δυνατότητες και να αποφύγουμε να υποπέσουμε στον πειρασμό να παίξουμε όλα τα χαρτιά μας ε, σε μία μόνο τεχνολογία. Όπως είπε ο κύριος Ντέιβις, ε, καταβάλαμε υπερβολικές προσπάθειες και ίσως επικεντρώσαμε όλοι μας την προσοχή και τις προσπάθειες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό στην πατρίδα μου δημιούργησε τεράστια προβλήματα και μεγάλα ελλείμματα. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά δυστυχώς έχει δημιουργηθεί ένα χάος με αντιδικίες ε, στα δικαστήρια και με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν τεράστια στις επιχορηγήσεις. Η μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων που αυτή τη στιγμή είναι το 80% της ε, φωτογενούς ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια διαδικασία χρονοβόρα. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης του διοξιδίου του άνθρακα είναι ένα, μια τεχνολογία που θα πρέπει να διερευνηθεί, να αξιοποιηθεί ώστε να μειώσουμε τα καυσαέρια χωρίς όμως ε, να αποποιηθούμε, να θυσιάσουμε τη χρήση των ορυκτών καυσίμων που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πηγή ενέργειας γιατί έχουν πιο ανταγωνιστικές τιμές. Η κυρία Φόρ, την οποία συγχαίρω για την ε, εξαιρετική της γραμμαδότηση που δεν μας ξαφνιάζει, ε, μας υπενθυμίζει λοιπόν στη γνωμοδότηση η κυρία Φόρτ ότι αν αρνηθούμε αυτή τη τεχνολογία να αποφύγουμε σοβαρές επενδύσεις στην τεχνολογία αυτή στα πλαίσια της μακροχρόνιας ενεργειακής μας στρατηγικής θα ε, εμποδίσει και τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές αλλά και τις παγκόσμιες προσπάθειες για την περιβαλλοντική πολιτική. Οπότε βρισκόμαστε σε μια στιγμή αποτελμάτωσης δυστυχώς των προγραμμάτων και στη γνωμοδότηση της κυρίας Φόρντ αλλά και ε, με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιστεύω ότι θα δοθούν ενάυσματα για να αναζωογονηθεί και πάλι μια προσπάθεια και μια τεχνολογία που φαίνεται είναι απαραίτητη. Ευχαριστώ κυρία Μαντουρέλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ένα σύντομο σχόλιο θα ήθελα να κάνω μόνο. Και εγώ πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να παρασυρθούμε σε μία λαθασμένη συζήτηση και το αν θα πρέπει ένα τμήμα των κονδυλίων για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια να το εφιερώσουμε στην τεχνολογία δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα. Εγώ πιστεύω ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να επιδιώξουμε την ανάπτυξη των αντίστοιχων τεχνολογιών για να μειώσουμε τι κλιματικέ αλλαγέ. Φυσικά εξαρτώμαστε από τα ορυκτά καύσιμα και η τεχνολογία αποθήκευση και δέσμευση του άνθρακα θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των καυσαίριων. Άλλωστε έχει γίνει μεγάλη προεργασία και πολλέ προσπάθειε. Ήδη έχουμε διάφορε τεχνολογίε στη διάθεσή μας για δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα και μπορούμε πια να περάσουμε σε φάση εφαρμογή σε επίδειξη τουλάχιστον αυτών των τεχνολογιών σε μεγάλη κλίμακα. Ε, βέβαια, τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ε, σε φάση που θα μπορούσαν να περάσουν σε αναπτυξιακό επίπεδο, αλλά διανύουν τεράστια προβλήματα ε, εν μέρη και μεταξύ της χαμηλής τιμής του άνθρακα στο σύστημα εμπορίας ε, ε, άνθρακα, στο ETS. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να πετύχουμε την απαραίτητη κινητοποίηση αυτού του προγράμματος. Είναι αξιέπινη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προτείνει ε, προτάσεις υποστήριξης του, της τεχνολογίας CCS. Αυτό είναι το πρώτο βήμα γιατί είναι σαφές ότι θα πρέπει να προτείνουμε νέα μέτρα πια, ώστε οι επιχειρήσεις ε, που θα αποφασίσουν να περάσουν σε σχέδια επίδειξης αυτής της τεχνολογίας ε, να έχουν, τύχουν κάποιες υποστήριξεις. Γι' αυτό και συμφωνώ με τις περισσότερες προτάσεις ηγετρίας. Και συμφωνώ και με τη σκιώδη ηγετρία και με τα σχόλια των ε, συναδέλφων. Δεν θα επαναλάβω λοιπόν τα προηγούμενα σχόλια. Συμφωνώ με τους συγητές. Συγγνώμη, Πρόεδρε, εάν θέλουμε να μειωθεί ο αντίκτυπος του διοξιδίου του άνθρακα στις, ε, στην κοινωνία μας, θα πρέπει να παράγεται λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα. Άρα θα πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη θέληση. Είμαστε υπέρ της τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει να δράσουμε ώστε να βρούμε τα χρηματοδοτικά μέσα, ώστε να, εφαρμοστεί, να εφαρμοστούν αυτές οι νέες τεχνολογίες και να βρεθούν και τα μέσα. Το διοξίδιο του άνθρακα όπως και το χρήμα ε, δεν είναι άοσμο. Γι' αυτό θα πρέπει ε, να δράσουμε άμεσα. Ε, ο άνθρακας... Un coup défiant το τα σχιστολιθικά αέρια μας το κατέδειξαν αυτό και βλέπουμε ότι μπορούμε να δαπανίσουμε πολύ άνθρακα για να παράγουμε περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια. Αν περιμένουμε το 2020 για να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια από διοξίδιο του άνθρακα, και να μολύνουμε περισσότερο τον ε, ορίζοντά μας, τότε δεν θα έχουμε καταφέρει ε, τίποτα. Έγινε λόγος για ιδιωτικοποίηση των κερδών και να αφήσουμε στον Ευρωπαίο φορολογούμενο να αντιμετωπίζει το όλο θέμα. Η Επιτροπή έχει το λόγο. Ποιος θα λάβει το λόγο από την Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο, όποιος την εκπροσωπεί για τρία λεπτά. Ελίνκα Μπάλαν από την Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, το πρώτο τμήμα. Σας ευχαριστώ που μας δώσατε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στη συζήτηση. Ε, έξι συμβάσεις έχουν υπογραφεί το 9 της τάξης του ενός ε, της και μόνο ένα, μία από τις τέσσερις συμβάσεις ε, τρέχει ακόμα. Ε, δύο δυστυχώς ακυρώθηκαν διότι υπήρξε ατελής μεταγραφή της οδηγίας CCS και αυτό ιδιαίτερα στη Γερμανία. Τα, οι τέσσερις άλλες συμβάσεις προχωρούν με ταχύς ρυθμούς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε επαφή με τους αναδόχους έτσι ώστε να ληφθούν αποφάσεις ε, για τις τελικές επενδύσεις. Για τις δύο συμβάσεις που έχουν ακυρωθεί και ιδιαίτερα για το σχέδιο της Γερμανίας, Βάτεν, έχει ληφθεί υπόψη ότι ότι υπήρξε κοινοποίηση αυτών των σχεδίων έτσι ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύστημα CCS. Δεν ταπανήθηκαν ε, όλα τα κονδύλια, αλλά τα προγράμματα αυτά μας βοήθησαν έτσι ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα το πρόγραμμα, το πρόγραμμα δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα. Ελπίζουμε να αποφασίσουμε για, το, για τις επενδύσεις, για τα τέσσερα υπολοιπόμενα προγράμματα και συμβάσεις. Θα δούμε πώς ε, είχε ο επιμερισμός των δαπανών και πόσα χρήματα θα δαπανηθούν για τις τέσσερις συμβάσεις και πόσα θα επιστραφούν στα κρατη διότι αυτό προβάλλει ο κανονισμός EPR. Ευχαριστούμε κυρία Φόρτ. Ευχαριστώ συνάδελφοι για τα πολύ σημαντικά θέματα που θίξατε. Σας ευχαριστώ γιατί μιλήσατε για μεγαλύτερη ε, δημόσια ενσυνειδητότητα. Μπορούμε να μάθουμε πολλά από την Νορβηγία η οποία ασχολείται με το θέμα του διοξιδίου του άνθρακα εδώ και 15 χρόνια, εκεί όπου υπήρχαν διαρροές. Και θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη αποθήκευση στις ανοιχτές θάλασσες. Και στον Καναδά οι εθνικές κυβερνήσεις ε, προσπαθούν να αναλάβουν αυτόν τον κίνδυνο και να τον διαχειριστούν ως προς την αποθήκευση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόντι γιατί μιλήσατε για την δέσμευση του, του φυτικού, ε, της φυτικής προέλευσης άνθρακα. Αν θέλουμε να προωθήσουμε τα ορυκτά καύσισμα και την αντιμετώπιση του διοξιδίου, τότε θα πρέπει να, έχουμε, να κάνουμε με σχέδια ευρεία κλίμακας για να βοηθήσουμε και τον βιομηχανικό τομέα. Ευχαριστώ, Κρίς, γιατί τόνισες ότι το κόστος έχει μειωθεί και το οποίο σημαίνει ότι το CCS μπορεί να είναι πιο αποδοτικό σε σχέση με τις ανανεώσιμες, διότι το κόστος είναι ύψης της σημασίας για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Γι' αυτό θα θέλαμε να έχουμε μια ουδέτερη τεχνολογία προσέγγιση. Μην ε, μειώσουμε την εμβέλεια της εργασίας για τον ορίζοντα 2020, διότι αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπίσουμε και το CCS. Αυτό μας απασχόλησε και στις τελικές μας συζητήσεις. Γι' αυτό ας ε, γίνει σωστή χρήση των χρημάτων. Ευχαριστούμε την Επιτροπή για την ενημέρωση. Θα ήθελα εκεί που υπάρχουν προσκόμματα σε αυτή την τεχνολογία να αρθούν. Και εάν το καταφέρουμε αυτό, δηλαδή να άρουμε τα προσκόμματα έτσι ώστε οι επενδυτές να προωθήσουν αυτά τα σχέδια, τότε θα έχουμε ανταποκριθεί στο ζητούμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σας υπενθυμίζω στους, υπενθυμίζω στους συναδέλφους ότι θα πρέπει να υποβληθούν οι τροπολογίες μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Περνάμε τώρα στην έκθεση ΟΔΙ και έχει το λόγο ο Ζαμπιέρ για την τεχνολογική και βιομηχανική βάση της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας παρουσιάζω μια γνωμοδότηση που εμπίπτει στο άρθρο 50 με την υπο... σε συνεργασία με την Υποεπιτροπή Άμυνας και την ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Γι' αυτό και είναι πολύ πεισμένο το χρονοδιάγραμμά μας, πολύ βραχή και σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες που καταβάλλατε κυρία Πρόεδρε με την Γραμματεία για να συνεδριάσουμε εκτάκτως και να ψηφίσουμε ώστε να διαβρύνουμε κάπως την προθεσμία μας για την κατάθεση των τροπολογιών. Την γνωμοδότηση την υποβάλλω στη συνεργασία με τον συνάδελφο Γκάλερ, που είναι ο εισηγητής γνωμοδότησης στην Υποεπιτροπή Άμυνας και ευχαριστώ και τους εισηγητές των υπόλοιπων πολιτικών ομάδων για τη συμβολή τους και γιατί έχουμε και γνωμοδότηση στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Εμείς θα ενδιαφερθούμε κυρίως ε, για τις βιομηχανικές πτυχές, ε, τις πτυχές της έρευνας και σε, μικρότερη, ε, σε μικρότερο βαθμό για την ενέργεια. Και φυσικά μιλούμε και για την βιομηχανική πολιτική για της, ε, το τομέα της άμυνας. Δυστυχώς εξαιτία των οικονομικών δυσκολιών των κρατών μελών και της λιτότητας ε, περιορίζονται και οι αμυντικοί προπολογισμοί. Θα πρέπει λοιπόν ως Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσουμε τους πόρους από κοινού ή να επιμερίσουμε τις δαπάνες μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Βανεροπόη που συγκάλεσε μια έκτακτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Δεκέμβριο και υπό αυτή την προοπτική υπό Επιτροπή Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκίνησε αυτό το διάβημα ε, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει όπως και έκανε τελικά μία ανακοίνωση για την ε, βιομηχανική βάση της άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις βιομηχανικές πτυχές πρώτα, τη βιομηχανική πολιτική, η γνωμοδότησή μου προτείνει να κρίνουμε ότι έχει έρθει η στιγμή να τεθεί τέρμα στον κατακαιρματισμό της αγοράς άμυνας, τόσο όσον αφορά τη ζήτηση και όσο αφορά και την προσφορά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κατακαιρματισμός που τον πληρώνουμε πολύ ακριβά οι αμυντικές συμβάσεις θα πρέπει να αναγνωριστούν ως ιδιαίτερες λόγω σχεδόν αποκλειστικά της κρατικής ζήτησης, της περιορισμένης προσφοράς και της μεγάλης εμπιστευτικότητας στις οποίες υπόκεινται αυτές οι συμβάσεις, οι αμυντικές συμβάσεις. Εν συνεχεία, προτείνω να θεωρήσουμε ότι η αμυντική βιομηχανία είναι επίσης ιδιαίτερη, λόγω τη υποχρέωση τη να αντιμετωπίσει μακρέ περιοδου ανάπτυξη και να διατηρεί συστήματα σε λειτουργία επί δεκαετίε, λόγω του σημαντικού και αυξανόμενου κόστου των προγραμμάτων, καθώ και λόγω τη έντονα ελεγχόμενη εμπορία των προϊόντων από την πλευρά των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Στηρίζουμε το, δικτό, το διτό χαρακτήρα των βιομηχανικών ικανοτήτων ασφάλεια και άμυνα, ιδίω στους τομεί του διαστήματο, τη θάλασσα και τη πολιτική αεροπορία. Και μάλιστα θα καταθέσω τροπολογία για να προσθέσουμε εδώ και τι τηλεπικοινωνίε Διαπιστώνουμε σήμερα ότι είναι ότι είναι προς το συμφέρον μας η ανάπτυξη του συστήματος Γαλιλαίο σε σχέση με τις ε, ε, κατασκοπευτικές ε, δραστηριότητες των ΗΠΑ και δεν θα πρέπει να εξαρτώμαστε από το σύστημα GPS, ιδιαίτερα αν διακόψουν το σήμα. Γι' αυτό καλούμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να στηρίξει την αμυντική βιομηχανική και τεχνολογική βάση που αποτελεί ιδιαιτερότητα ορισμένων εξοπλισμών για τους οποίους θα πρέπει να διατηρηθεί μια στρατηγική αυτονομία και μια επιχειρηματική, επιχειρησιακή κυριαρχία. Ένα θέμα που θα συζητηθεί σίγουρα και περιμένω εδώ με ανυπομονησία της απόψης των πολιτικών ομάδων και των εθνικών αντιπροσωπιών είναι ε, η ιδιαίτερη θέση που θα μπορούσαν να έχουν οι ευρωπαϊκοί οικονομικοί φορείς στον τομέα της άμυνας και κυρίως τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν που θα συζητήσουμε και σε πολιτικό επίπεδο και τα οποία σχετίζονται με την απασχόληση, με τους τόπους απόφασης και παραγωγής του ευρωπαϊκό έδαφος, ώστε να καθίσετε δυνατή η προστασία των τόπων αυτών, γιατί η ιστορία μας έχει δάξει ότι κάθε φορά που γίνεται επίθεση ενός μιας περιοχής, αυτές, αυτοί οι τόποι είναι πολύ ευάλωτες επιθέσεις, γι' αυτό και θα πρέπει να προστατεύσουμε την αμυντική μας βιομηχανία, και σε επίπεδο ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αλλά και ε, στην πράξη. Επίσης στηρίζουμε την Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Έχουμε παράγραφο για το διάστημα που διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στον τομέα της άμυνας και έχουμε και πολλές παραγράφους για την ασφάλεια την ηλεκτρονική, για να είμαστε λιγότερο ευάλωτοι απέναντι στις επιθέσεις ε, που ίσω αντιμετωπίσουμε. Έχουμε και παραγράφου για τη συνεργασία στον τομέα τη διαλειτουργικότητας, δύο παραγράφου και για τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού αμυντικού υλικού και τέλος στηρίζουμε, απροτείνουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κάνουμε συστήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συνήθω κάνουμε στάσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά στην περίπτωση αυτή η γνωμοδότησή μας θα επιδοθεί στην Υποεπιτροπή Άμυνα και στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εγκρίνει ψήφισμα που θα δοθεί στο, Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Εκεί ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, χωρί να μειχθεί στο νομοθετικό επίπεδο, να δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι απαραίτητε οθήσει και να καθορίσει του προσανατολισμού και τι γενικέ πολιτικέ προτεραιότητε για την ενίσχυση τη αμυντική, βιομηχανική και τεχνολογική βάση. Τέλο, κυρία Πρόεδρε, για να μην χρονοτριβήσω, θα ήθελα να αφαιρθώ στα δημοσιονομικά θέματα θα ήθελα να αφήσουμε κατά μέρο αυτή τη στιγμή τα ζητήματα του προπολογισμού, γιατί είχαμε κάποιε δύσκολε συμφωνίε για τον ορίζοντα του 2020 και θα δούμε ίσω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου παραπέμψει στις αποφάσεις των πολιτικών ομάδων σε ό,τι αφορά τις ευρωεκλογές του 2014 και στη ρήτρα αναθεώρησης του δημοσιονομικού πλαισίου του 2016. Θα δούμε. Ίσως τότε συμφωνήσουμε και για τα επιμέρους δημοσιονομικά σκέλη αυτής της πρότασης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο ε, Οντί. Το... κύριο Γκέρεκ. Ευχαριστώ. Ε, η αμυντική κατάσταση στην Ευρώπη κυρίως η αποχώρηση του Αμερικανικού στρατού και κάποιες ε, ταραχές σε τρίτες χώρες, Αίγυπτο, Συρία, πρόσφατα και προηγουμένως και στη Λιβύη, όλα, όλα αυτά τα γεγονότα θα πρέπει να μας οδηγήσουν να ενισχύσουμε τη, την τεχνολογική μας και αμυντική βάση στην Ευρώπη. Υπάρχουν τέσσερις ε, λόγοι που επηρεάζουν και απειλούν την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική ασφάλεια, υπάρχει κίνδυνος Υπάρχει κίνδυνος και από τις τρίχες χώρες που έχουν ε, πυράβλους ε, μέσα ή ε, μεγάλες εμβέλειας, μέσου ή μεγάλου βεληνικούς. Επίσης, τι γίνεται με τις εγκαταστάσεις σε χώρες όπως το Μαλί ή με απειλές τρομοκρατικού χαρακτήρα. Επίσης μπορούμε να υποστούμε απειλές όχι μόνο από αέρος αλλά και από ξηράς και θαλάσσης. Γι' αυτό χρειαζόμαστε να εναρμονίσουμε τις, προστά... τις προσπάθειες των χωρών μελών προκειμένου να ενισχυθεί το, το επίπεδο ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την βιομηχανική, τεχνολογική και αμυντική μας βάση. Πολύ σημαντικές είναι οι έρευνες, ε, οι στρατιωτικές για τα θέματα της ασφάλειας, αλλά δεν μπορούν να δοθούν ε, δημόσια τα αποτελέσματά τους. Θα πρέπει να δούμε κάποια στήματα διάγνωσης, ε, διαστημικής πλοήγησης, ε, ραντάρ, πολύ πιο συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, ίσως δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αντιπυραυλικής ασπίδας. Και επίσης υπάρχουν και νομικά θέματα ενοποίησης και εναρμόνισης σε θέματα χρησιμοποίησης οχημάτων ε, ξηράς ε, και ε, ροσκαφών, αλλά και φυσικά εναρμόνιση των πυρομαχικών, ώστε να χρησιμοποιούνται τα ίδια πυρομαχικά να μπορούν να χρησιμοποιούνται σε εξοπλισμούς διαφόρων χωρών. Θα πρέπει επίσης να ζητήσουμε μεγαλύτερη εξειδίκευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγαλύτερη συνέργεια προκειμένου να δημιουργηθεί ενίσχυση του αμυντικού δυναμικού και των μεμονωμένων χωρών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, όπως έγινε και στο ΝΑΤΟ, ε, τα, τα, οι αμυντικές ταπάνες θα πρέπει να ανέρχονται στο 2% του εθνικού ΑΕΠ. Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα πλαίσιο, γιατί εκεί υπάρχει πρόβλημα, όπως είπε ο κύριος Σοντή, ε, για τα απορίσματα αυτά των εξαιρετικά εμπιστευτικών ε, ερευνών της αμυντικής βιομηχανίας, θεωρώ ότι θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο χρειαζόμαστε ένα Ινστιτούτου στυλ Κοινού Κέντρου Ερευνών που θα ασχοληθεί με τα θέματα των αμυντικών εξοπλισμών και θα τη χάνει ε, ανεξάρτητης χρηματοδότησης από τον ορίζοντα το 2020 και φυσικά οι εργασίες ενός τέτοιου Ινστιτούτου θα πρέπει να είναι απολύτως εμπιστευτικές και μυστικές. Ευχαριστώ. Κύριος Πρόντι. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα λεπτό. Έχω την εντύπωση ότι στην ουσία Έχουμε να κάνουμε με μια διακυβερνητική διαχείριση της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής όπου επικαλύπτουν τα μεμονωμένα συμφέροντα των ε, κρατών μελών των όλο τομέα. Αυτή η βιομηχανία άμυνας εξαρτάται από μία θαραλέα απόφαση, δηλαδή να έχουμε μία ευρωπαϊκή κοινή πολιτική άμυνας. Αν δεν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα, θα αναρωτιόμαστε συνέχεια γιατί δεν τα καταφέραμε στον ε, τομέα της άμυνας όπως τα καταφέραμε στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας. Έχουμε να κάνουμε με ένα επίπεδο παγκόσμιου ανταγωνισμού και εάν ήμασταν αποφασισμένοι η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί και να καλύψει και τη βιομηχανία άμυνας. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα με μια προσέγγιση άναντι, έτσι ώστε να έχουμε μια κοινή πολιτική άμυνας. Ευχαριστούμε η Επιτροπή. Δεν ξέρω κατά πόσο κάποιος θα ήθελε το λόγο. Έχετε το λόγο. Απλώς ε, θα ήθελα να μιλήσω εντάχει για να τονίσω τη σημασία αυτού του ζητήματος και την ε, αντίδραση του Κοινοβουλίου σε αυτή την ανακοίνωση καθώς ε, εν μάλλον του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Εάν θέλουμε να επιτελεστεί πρόοδος σε αυτό τον τομέα, στον τομέα της άμυνας, θα πρέπει να γίνει μια συλλογική προσπάθεια και από τα τρία θεσμικά όργανα, τα κράτη-μέλη και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, ε, ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Βιομηχανίας Άμυνας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Οντί έχει το λόγο και πάλι. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο συναδέλφους που έλαβαν το λόγο και που υποστήριξαν τη βασική αυτή ιδέα, η πολύ καλή ιδέα να δημιουργηθεί ένα κοινό κέντρο ερευνών στον τομέα της άμυνας ε, με μια διευρυμένη εντολή και ευχαριστώ τον συνάδελφο Πρόντι. Δεν πρόκειται για θέματα πολιτικής θέλησης, αλλά πρόκειται για έναν ευαίσθητο τομέα γιατί μιλάμε για θέματα εθνικής κυριαρχίας. Νομίζω ότι μέσα στα πλαίσια των αλλαγών στο, σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει και η Ευρώπη να υπερασπίσει τι τον εαυτό της και να υπερασπιστούμε τις αξίες και τις ιδέες οι οποίες μας διέπουν. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω με τις τροπολογίες να φτάσουμε σε συμβιβασμούς που θα προβάλλουμε στην Υποεπιτροπή Άμυνας. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που με βοήθησαν καθώς και τους συνεργάτες μου για την εκπόνηση αυτού του σχεδίου νομοδότησης. Ωραία, ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο Όντι. Πριν περάσουμε στις ψηφοφορίες, θα ήθελα να ε, τονίσω κάτι που ζητήθηκε ως προς τη δυνατότητα να ψηφίσουμε στο Στρασβούργο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο για τις τροπολογίες όπως γνωρίζετε, αυτό σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα των αιθουσών. Βρήκαμε μία αιθούσα, η οποία όμως δεν είναι και η καλύτερη για τις ανάγκες μας. Δεν υπάρχει επαρκής χώρος, γι' αυτό θα ήθελα να αφήσουμε ανοιχτό αυτό το ζήτημα και η γραμματεία θα μας πληροφορήσει εν καιρό. για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε αίθουσα στη διάθεσή μας για τις 7 Οκτωβρίου. Και έτσι θα ε, δούμε κατά πόσο πρέπει να κρατήσουμε ή όχι την αρχική ημερομηνία υποβολής τροπολογιών. Μέχρι αύριο θα μας έχει απαντήσει η γραμματεία. Σας ευχαριστώ ναι. πολύ. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες.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 Ας κάνουμε μία δοκιμή. Ελπίζω να περάσατε ένα καλό καλοκαίρι. Ερώτηση ήταν αυτή και ελπίζω να απαντήσετε όλοι θετικά. Γίνεται μία δοκιμή για να δούμε αν λειτουργεί το σύστημα, οι κάρτες μας. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Πέρασε. 31 υπέρ, 3 κατά και 4 ε, αποχές. Μπουτιχόφερ. Περνάμε στην έκθεση. Κυρία Πρόεδρε, λυπούμε, αλλά έχω ξεχάσει την ε, κάρτα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Σας παρακαλώ, μην με ξεχνάτε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ τη συνάδελφα Μαντουρέλ. Θα το λάβουμε υπόψη. Ε, ζητήθηκε να ψηφίσουμε en bloc τα πρώτα σημεία που αφορούν τον προϋπολογισμό γιατί σχετίζονται με την έγκριση του ιδίου. Εάν συμφωνείτε λοιπόν, Ψηφίζουμε on block όλες τις τροπολογίες που αφορούν ε, το τμήμα Restored Budget. Δέχεστε όλοι αυτό το μπλοκ υπέρ. Κατά. Ένας αποχές. Ωραία. Εγκρίνονται οι τροπολογίες αυτές. Περνάμε τώρα στην Ήτρε 01 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, ε, ας γίνει έλεγχος καλύτερα. Αρχίζει η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Πέρας. 19 υπέρ, 20 κατά, 2 αποχές ε, απορρίπτεται. Ήτρε 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 02 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται 36 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται 37 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 04. Άμε συγχωρείτε, λέει πρόεδρος. 03. Υπέρ. Όχι. Ψηφίσαμε την 81. Τώρα ψηφίζουμε την Ήτρε 5903. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 04 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία, 04 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 29 υπέρ, 12 κατά εγκρίνεται. 06 υπέρ, κατά. Δεν είναι απόλυτα σαφές. Ήταν 4 υπέρ, κατά. Ε, δεν μου πήγε καλά το καλοκαίρι, δεν ε, μπορώ να προχωρήσω με τη δέουσα ταχύτητα. 06, 06 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ, κόντρο, κατά, αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 09 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ, κατά αποχές ας επαληθέψουμε. 78 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας 7 υπέρ, 33 κατά. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 77 στο 70, 73 αρχίζει η ψηφοφορία, επαληθεύουμε. Πέρας. 37 υπέρ, 5 κατά, εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 32 υπέρ, 2 κατά, 8 αποχές ε, εγκρίνεται. Να συγχαρούμε τον εισηγητή. Έχουμε τώρα μία ε, έκθεση νομοθετικού περιεχομένου για το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης. Ψηφίζουμε την ε, έκθεση νομοδότησης. Αρχίζει η ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 40 υπέρ, 1 κατά, καμία αποχή. Σας ευχαριστώ, ζητώ συγγνώμη γιατί κάθε αρχή και δύσκολη. Περνάμε στα επόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης τώρα. Εάν κάποιος θέλει να φύγει από την αίθουσα, να φύγει άμεσα παρακαλώ για να μας επιτρέψει να συνεχίσουμε. Marianne, Ωραία. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Έχουμε αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Γι' αυτό σας παρακαλώ να προχωρήσουμε. Έκθεση Βαλεάν. Η συνάδελφος Βαλεάν δεν είναι παρούσα. Ε, ο συνάδελφος Κρόιτσμαν θα παρέμβει εξ ονόματός της. Ευχαριστώ. Και στο όνομα της κυρίας Βαλεάν που είναι απούσα λίγες ιδέες για την έκθεσή της. Περίπου 60 τροπολογίες. Από μια πρώτη ανάλυση δεν βλέπει να υπάρχουν σημαντικές διαστάσεις ε, απόψεων ανάμεσα στους στόχους και στα μέσα. Πρέπει να δοθούν επενδύσεις για την υποδομή ενέργειας, οι πληροφορίες που δίνουν οι εταιρείε να είναι εμπιστευτικές. Η κυρία Βαλεάν προτείνει συμβαστικές τροπολογίες για τα εκρεμή θέματα, όσο το δυνατόν συντομότερα, αλλά τονίζει προς την κατεύθυνση των συναδέλφων ότι το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ στενό και ελπίζει να μπορέσουμε να συνεργαστούμε σύντομα ώστε να καταλήξουμε σε συμφωνία εντός δύο εβδομάδων πριν από την, τροπολογία, ε, πριν από την ψηφοφορία συγγνώμη, που προβλέπει για τις 18 ενάτου. Κυρίως τρία θέματα. Πρώτον, πότε θα πρέπει να γίνεται η κοινοποίηση για την τροπολογία 39, 26 κτλ. Εκεί υπάρχουν ορισμένε ανησυχίες εάν η κοινοποίηση γίνεται υπερβολικά πρόημα διότι αυτό ίσως προκαλέσει τον κίνδυνο να διακυβευτούν ορισμένες εμπιστευτικές πληροφορίες. Ωστόσο, εάν οι κοινοποίησεις γίνουν μόνο για τα κτίρια, αυτό θα μειώσει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Τα δεκαετή σχέδια ανάπτυξης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με και χωρίς τις τελικές αποφάσεις και τις επενδύσεις σε συνεργασία με, τις, με την Κομισιόν θα πρέπει να γίνει ε, καλύτερη διατύπωση για την ε, ταυτοποίηση των δεδομένων για να αποφεύγεται η διπλή κοινοποίηση και η Κομισιόν να δώσει τη σωστή, τους σωστούς τύπους για τις χώρες μέλη και για τα άλλα δεδομένα, ώστε να μην χρειάζεται να αποφασίζουν ποιες πληροφορίες ήδη έχουν δοθεί για να αποφευθεί σύγχυση και αποφυγή ευθυνών. Θα πρέπει να καταλήξουμε μεταξύ μας και σε συμβαστική λύση για τις κατηγορίες που θέλουμε να περιλάβουμε στο επίπεδο εφαρμογή και στα παραρτήματα. Ορισμένοι συνάδελφοι έχουν προτείνει τροπολογίες για την τροποποίηση των κατηγοριών των εγκαταστάσεων. Πρέπει να εξετάσουμε την εφαρμοσιμότητα αν οι χώρες μέλη δηλαδή μπορούν όντω να συλλέγουν τα δεδομένα αυτά, έχοντας υπόψη και την ανάγκη ελαχιστοποίησης του γραφειοκρατικού βάρους. Η κυρία Βαλεάν θεωρεί ότι έχει νόημα για ορισμένες κατηγορίες ανανεώσιμων να ε, εξεταστεί αν υπάρχουν τα δεδομένα αυτά. Κατά τα άλλα, θεωρεί ότι μπορούν να συζητηθούν τα υπόλοιπα θέματα στις ε, συναντήσεις των σκιωδών. Υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει, αλλά πιστεύει ότι μπορούν όλα αυτά να συζητηθούν εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και αναμένει την περαιτέρω συνεργασία και των άλλων ε, σκιωδών εισηγητών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βρίσκω καλή την έκθεση της κυρίας Βαλεάν, ο κύριος Λάνγκεν. Οι τροπολογίες εν μέρη δέχονται την έκθεση, εν μέρη αποσκοπούν σε μια αποδυνάμωσή της. Ακόμα δεν έχουμε τις συμβαστικές τροπολογίες της κυρίας Βαλεάν που θα μας επιτρέψει να κρίνουμε καλύτερα. Είναι 61 οι τροπολογίες και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και ορισμένες που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση όλου του εγχείρηματο. Για παράδειγμα, ο κύριος Στάσεν, Ολλανδός, σε πολλές τροπολογίες του ζητεί η μεταβίβαση των δεδομένων να γίνεται μοναχά σε εθελοντική βάση. Εγώ δεν το θεωρώ σκόπιμο αυτό. Εάν υπάρχει, αν γίνεται η διαβίβαση των δεδομένων για τις υποδομές ενέργειας θα πρέπει αυτό να προσφέρει και κάποια προστιθέμενη αξία. Ο κ. Ζαντό εξάλλου περιλαμβάνει εκτός από τον άνθρακα και, άλλου, και άλλα είδη ενέργειας που χρησιμοποιούνται και στις μεταφορές και ζητεί και για αυτά να δίνονται τα σχετικά δεδομένα και ορίζει στο άρθρο 2 εγκαταστάσεις οι οποίες δεν, δεν ε, αναφέρονται σε κανένα άλλο σημείο. Εκτός από τις οποίες της κυρίας Στάσεν νομίζω ότι μπορούμε να εγκρίνουμε τις συμβαστικές τροπολογίες ταχύτατα, γιατί είμαστε σύμφωνοι σε μεγάλο βαθμό. Το θέμα που τίθεται ως κριτήριο είναι από ποιο μέγεθος και πάνω θα είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των δεδομένων, αν θα είναι για μεμονωμένες εγκαταστάσεις ή όχι. Αυτά όμως όλα είναι δυνατόν να συζητηθούν. Βρίσκω να είναι θετική η βάση έτσι ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα σε μια ε, συμφωνία. Κορέρα το κάμπος. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βαλεάν για την εργασία της και τις τροπολογίες των συναδέλφων, διότι συμφωνούμε με τις ε, τροπολογίες των ε, συναδέλφων θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής σε σχέση με τα επενδυτικά επενδυτικά σχέδια στην ενεργειακή υποδομή και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το υγροποιημένο αέριο καθώς και τα σημεία διασύνδεσης. Θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν επικαλύψεις ως προς την υποχρέωση ε, κοινοποίησης, έτσι ώστε να μην επιβαρύνουμε τη γραφειοκρατία. Συμφωνούμε με τις τροπολογίες οι οποίες ε, καλύπτουν τον ενεργειακό τομέα, την Euratom, τις υποδομές και ούτω καθεξής. Επίσης δεν θα πρέπει να υπάρξει ε, αλόγιστος διοικητικός ε, φόρτος, ιδιαίτερα ε, ως προς τα κατόφλια ικανότητας παραγωγής. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα έργα τα οποία έχουν τύχει αδειοδότησης και να εντάξουμε όλα τα σχέδια σε μια διαδικασία κοινοποίησης για να υπάρξουν οι κατάλληλες επενδύσεις με βάση την αναγνώριση των χασμάτων που υπάρχουν και την αποκατάσταση των ενεργειακών αναγκών. Από την άλλη πλευρά θεωρούμε ότι η πρόταση Επιτροπής διασφαλίζει όλα τα μέτρα, εξασφαλίζει όλα τα μέτρα ε, για την ε, διατήρηση της εμπιστευτικότητας, αλλά ορισμένες τροπολογίες είναι υπερβολικές σε σχέση με το μέλημα αυτό. Είμαστε στη διάθεσή σας για να συνεργαστούμε και παρά το περιορισμένο χρόνο νομίζω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια αίσια έκβαση σύντομα. Ζαντό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Ε, είναι ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο το οποίο επεξεργαζόμαστε εδώ και χρόνια. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε μια τεκμηριωμένη άποψη και μια, να κάνουμε μια πλήρη επισκόπηση του ενεργειακού τοπίου. Γι' αυτό και συμφωνούμε με την εισηγητρία ότι για τον άνθρακα ότι όλα τα δικαιωμένα στον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα μας ε, δημιουργήσουν μια πλήρη επισκόπηση της κατάστασης. Επίσης ε, θα θέλαμε τα κατώτατα όρια εφαρμογής να μειωθούν ε, περαιτέρω. 5 MW ΜΒ προτείνει για τα αιωλικά πάρκα ε, η συγκήτρια. Εμείς πιστεύουμε ότι από τα 10 ΜΒ στο 1 ΜΒ θα πρέπει να μειωθούν και τα κατώτατα όρια για τα φωτοβολταϊκά. Δεν θεωρούμε αντίθετα και πολύ ρεαλιστικό, θα το συζητήσουμε όμως με την εισηγήτρια, το θέμα της ένταξη των υποδομών σε τρίτε χώρε, ακόμη και αν υπάρχει μια διασύνδεση με χώρε μέλη. Και θα υπάρξει πρόβλημα εφαρμογή για ένα τέτοιο μέτρο. Επίσης, θα θέλαμε στο πρόγραμμα να συμπεριληφθεί μείωση της ε, κατανάλωση ενέργειας, πληροφορίες ε, για διάφορες ε, τεχνολογίες, το θέμα της αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων και επίσης ε, πληροφορίες για τα δίκτυα άθρακα και για τα θέματα παραγωγής ε, θερμότητας. Θέλουμε περισσότερη διαφάνεια και μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών. Ευχαριστώ και θα υποβάλουμε τροπολογίες επίσης. Ε, Ευχαριστώ. Αναφίβολα, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τα παιδικά σχέδια σε σημαντικές ενεργειακές υποδομές ε, μας επιτρέπει μια καλύτερη συνολική ανάλυση και επισκόπηση του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος και σίγουρα ε, είναι στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών. Δύο όμως σημεία θα πρέπει να τέχουν ιδιαίτερης προσοχής γιατί ίσως δημιουργήσουν προβλήματα και δεν είναι τυχαίο που υποβλήθηκαν τόσες τροπολογίες για τα σημεία αυτά. Ένα από τα δύο σημεία είναι ότι θα πρέπει να αποφύγουμε την ε, επιβολή υπερβολικού γραφειοκρατικού άχθους ή διοικητικού άχθους στις εθνικέ αρχές. Και δεύτερο θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι αφορά τι ε, εμπορικά ευαίσθητε πληροφορίε. Άλλο σημείο που επισήμανε η συγκεντριά για βελτίωση είναι η ανάγκη της συμπερίληψης των υποδομών του άνθρακα στο πεδίο εφαρμογής ε, του κανονισμού αυτού. Είναι αλήθεια ότι οι επενδύσεις αυτές είναι ε, μικρότερες από άλλες, αλλά θα πρέπει να υπόκεινται στην ίδια υποχρέωση κοινοποίηση. Αλλιώς ε, δεν θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκεντρώσει ακριβείς πληροφορίες και Γι' αυτό και τέτοιες ελληνικέ πληροφορίες ε, θα ήταν άχρηστες. Επίσης, οι πληροφορίες ε, που θα κοινοποιούνται θα πρέπει να ε, υπόκεινται σε ανάλυση όχι μόνο για στατιστικές μελέτες, αλλά προκειμένου να, γίνουν, να υποβληθούν στη συνέχεια συγκεκριμένες προτάσεις. Μόνο έτσι έχει νόημα μια ανάλυση των διαφόρων στοιχείων. Και Πιο συγκεκριμένα, μιλάει εδώ ένα Ισπανό και φαντάζομαι θα συμφωνήσουν και οι Πορτογάλοι. Χρειαζόμαστε τέτοιε πληροφορίε για να εντοπίσουμε ε, κενά και αδυναμίες ε, και ελλείψεις που υπάρχουν μερικές φορές στις ε, διαμεθοριακές διασυνδέσεις. Γιατί αν δεν διορθωθούν αυτές οι αδυναμίες δεν θα μπορέσουμε καν να μιλάμε για εσωτερική αγορά ενέργειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή ήδη έχει μελετήσει τις τροπολογίες και συμφωνούμε με ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με διασαφήσεις ως το πεδίο εμφαρμογής που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα και να μην υπάρχει επικάλυψη από διάφορες πηγές. Υπ' αυτή την έννοια οι τροπολογίες διασάφησης είναι πρόσδεκτες. Ως προς τα τρία σημεία που ανέφερε ο εισηγητής ή η εισηγήτρια, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι επενδύσεις. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε τα προγράμματα όπου έχουν ληφθεί αποφάσεις περί επενδύσεων ή να προχωρήσουμε παραπέρα ε, περιλαμβάνοντας και τα σχέδια που δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση ε, επενδυτικής υφήσης. Ως προς το δεύτερο βασικό σημείο που προαναφέρθηκε, να μην υπάρχει επικάλυψη ή διπλή κοινοποίηση, ε, εμείς ασχοληθήκαμε, μάλλον δώσαμε τελική μορφή το Νοέμβριο του 12 για την κοινοποίηση, διαδικασία κοινοποίησης υποδομών και ορίσαμε τομείς που καλύπτονται από άλλους τομείς και πηγές για να μην υπάρχει διπλή κοινοποίηση. Και έγινε και σύγκριση δεδομένων. Εάν λοιπόν θέλουμε να ξέρουμε τι χρειάζεται από τα κράτη-μέλη και τι μπορούμε να λάβουμε από άλλες πηγές, θα μπορούσαμε να καταβάλουμε μια προσπάθεια σε αυτό το τομέα. Ως προς τις ανανεώσιμες βεβαίως ε, οι μικρές πηγές ανανεωσίμων δεν καλύπτονται από αυτό τον κανονισμό και γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ως προς ανανεώσιμες ε, ε, μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας κοινοποίησης μη. Θα πρέπει να δούμε τι προϋπάρχει στα κράτη-μέλη για τις μικρές εγκαταστάσεις έτσι ώστε να τις συμπεριλάβουμε, αλλά αν δεν προϋπάρχουν θα είναι πολύ δύσκολη η συμπερίληψη. Ε, ως προς την τροπολογία για το πεδίο εφαρμογής, ε, υποβλήθηκαν μερικές τροπολογίες, θεωρούμε ότι ο κανονισμός καλύπτει το, την ηλεκτρική ενέργεια από άνθρακα και λιγνίτη, ε, κινητοποίηση στην συμπαραγωγή θέρμανσης και ηλεκτρισμού ήδη καταγράφονται στα παραρτήματα και αυτό αφορά και τα βιοκαύσιμα και τις σχετικές επενδύσεις. Δεν καλύπτεται η εξόριξη άνθρακα αυτά τα επενδυτικά σχέδια. Όμως θα πρέπει να, ίσως να περιμένουμε την αναθεώρηση που αναμένεται πριν από τα τέλη του 2016 και ενδεχομένως να συμπεριλάβουμε και άλλες πηγές. Η Επιτροπή είναι ευτυχής και προσβλέπει στις τροπολογίες συμβιβασμού για να συνεχιστεί η συζήτηση. Ευχαριστούμε. Κρόιτσμαν. Αν θέλει να αναφέρει κάτι ο κύριος Κρόιτσμαν. Στις 18 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Ήτρε. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα τη συναδέλφου Νίμπλερ. που αντικαθίσταται από τη συνάδελφο Χέλλερ, τον συνάδελφο. Ευχαριστώ θα διαπιστώσατε κι εσείς ότι δεν είμαι η κυρία Νίπλερ, η οποία όμως είχε μια άλλη ανηλυμένη υποχρέωση σήμερα και γι' αυτό με παρακάλεσε να τα πω εγώ. Το ιστορικό είναι γνωστό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική. Η κυρία Νίμπλερ ευχαριστεί και την Κομισιόν για τη συνεργασία, για την ανακοίνωσή της, δηλαδή της 28 Φεβρουαρίου. Τονίζει ότι στον διαστημικό κλάδο εργάζονται μόνο εντός εισαγωγικών 34.000 ε, επιστήμονες υψηλών ειδικών προσόντων τα όσα διδάγματα αντλούνται από την δραστηριότητα αυτή δεν καταλήγουν συνήθως μέχρι τον πολίτη. Παρόλα, αυτό, παρόλα αυτά είναι σημαντικά. Για παράδειγμα η τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας, διάφορα συστήματα ε, πλοήγησης. Ε, η Γεωργία επίσης επωφελείται πολύ από τις ε, γνώσεις που αποκτώνται από τη διαστημική έρευνα. Στην ανακοίνωσή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει η διαστημική πολιτική να περιοριστεί σε πέντε σημαντικούς στόχους που δεν θα αναφέρω, για την επίτευξη των στόχων αυτών προτείνει η Κομισιόν 37 επιμέρους μέτρα σε διαφόρους τομείς. Η εισηγήτρια κρίνει ότι εδώ θα πρέπει να μπουν κάποιες προτεραιότητες. Το σχέδιο εκθεσός τη, περιλαμβάνει 7 τομείς που θα πρέπει να απασχολήσουν ιδιαίτερα. Τα θεσμικά θέματα, Γαλλίος Κοπέρνικος, την διαστημική έρευνα ως ε, μοχλό ανάπτυξης, τον ρόλο της ανάπτυξης και της έρευνας, την επικοινωνία μέσω δορυφόρων και την ε, διαστημική έρευνα. Θα, αναφερθώ με λίγα λόγια στους διαφόρους τομείς για την θεσμική πτυχή. Εκεί μπαίνει η συνεργασία μεταξύ ESA, χωρών μελών κλπ. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι εδώ υπάρχει μεγάλος χώρος βελτίωσης της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή δηλαδή, Υπηρεσία Διαστήματος που θα πρέπει να αναλάβει το ιδιαίτερο ε, βάρος. Δεύτερο, για Γαλιλαίο και GMS που είναι οι εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Διαστημικής ε, Έρευνας πρέπει να δοθεί σημαντική προτεραιότητα, βελτίωση της επικοινωνίας εκμετάλλευση των πλονεκτημάτων του Γαλιλαίου και καλύτερη μεταφορά επικοινωνιακά. Τρίτο, ως μοχλός ανάπτυξης. Ασφαλώς το μέγα θέμα εδώ είναι η χρηματοδότηση. Πρόκειται για βιομηχανία υψηλών επενδύσεων με πολύ μακροχρόνιες αποσβέσεις. Οι επιχειρήσεις διστάζουν να επενδύσουν πολλά χρήματα διότι δεν είναι βέβαιο εάν θα βρεθούν πελάτες για τα προϊόντα που θα προκύψουν από την οικονομική αυτή δραστηριότητα. Πρέπει να ενισχυθεί με επιδοτήσεις διότι ιδίω ο τομέα της ρομποτικής μπορεί να ε, ενισχυθεί πολύ. Και επίσης η διαγωνιμοποίηση, cross-fertilization, δηλαδή μεταξύ διαφόρων τομέων, μπορεί να ωφελήσει πολλούς από αυτούς για την ανάπτυξη τεχνολογιών και επίσης πρέπει να εξετάσουμε και το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται η Ευρωπαϊκή Διαστημική Έρευνα. και που χρηματοδοτείται βέβαια κυρίως από τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Πρόσβαση στο διάστημα είναι το τέταρτο. Σημαντικό είναι εδώ να ανοίξουν αγορές άλλων χωρών μέσα από εμπορικές συμφωνίες, να δημιουργηθεί ανταγωνισμός με ίσους όρους, να υπάρχει ανεξάρτητη πρόσβαση στο διάστημα, γιατί αυτά είναι σημαντικά. Και στις προϋποθέσεις για την επιτυχία της βιομηχανικής πολιτικής. Πέμπτο, για το ρόλο της έρευνας και ανάπτυξης. Εδώ χρειάζεται βελτίωση του συντονισμού μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, ESA και χωρών μελών στα πλαίσια ενός χρονοδιάγραμματος μέχρι το 2020, καθώς και η αποφυγή επικαλύψεων. Τα προκύπτοντα δεδομένα θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο καλύτερης εμπορικής εκμετάλλευσης. Το έκτο, επικοινωνία μέσω δορυφόρων που παίζει πρωταρχικό ρόλο στην διαστημική βιομηχανία μπορούν οι, μπορούν οι δορυφόροι να χρησιμοποιηθούν και για το ευρέω φάσματο διαδίκτυο για να καλύψουν δηλαδή τι ανάγκε όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν θα πρέπει λοιπόν να εξετάσει τι μελλοντικέ ανάγκε δορυφορικών επικοινωνιών και στην επόμενη παγκόσμια διάσκεψη να φροντίσει ώστε να προστατευτούν τα δικαιώματα και συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δορυφορική επικοινωνία θα πρέπει να ληφθεί περισσότερο υπόψη μέσα στα πλαίσια της διαστημικής έρευνας από ό,τι γίνεται μέχρι τώρα στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, στο έβδομο θέμα για τα απορρίμματα στο διάστημα, το ερώτημα που τίθεται είναι σε ποιον ανήκει το διάστημα. Η συγγήτρια θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει ένα είδος παγκόσμιας διαχείρισης, global governance του θέματος αυτού και με πρόγραμμα για την υποστήριξη της παρακολούθησης του περιβάλλοντος που πρέπει να θεσπιστεί το δυνατόν συντομότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να εξασφαλιστεί και μια ανεξαρτησία από τις Ενωμένες Πολιτείες ιδίως σε ό,τι αφορά μια έγκαιρη προειδοποίηση για τους κινδύνους συγκρούσεων. 4 Σεπτεμβρίου η προθεσμία προπολογιών, 26 Σεπτεμβρίου η ψηφοφορία και Νοέμβριος 13 η ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκλάντε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την ε, ανάπτυξη της εκθέσεως του κυρίου Νίβλερ, κύριε Έλερ. Συνολικά, συμφωνώ με το περιεχόμενο της εκθέσεως Νίπλερ. Τονίζω ορισμένα πράγματα. Η ανακοίνωση της Επιτροπής είναι σημαντική, αλλά είναι και αμφισβητούμενη. γνωρίζω ότι θα υπάρξει διαφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιών από τη μια μεριά και χώρων μελών από την άλλη. Εμείς θα πρέπει εδώ να καταλήξουμε σε μια ομόφωνη τοποθέτηση και μετά να τη διαπραγματευτούμε με τις χώρες μέλη. Προσοχή να αποφύγουμε την επικάλυψη προσπαθειών. Ταυτόχρονα πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να συνδυάσουμε τις προσπάθειες, συνέργεια δηλαδή. Υπάρχουν καλές συνεργασίες, υπάρχουν καλές κοινοπραξίες, ας το πω έτσι. Αυτό θα είναι όμως, εδώ θα εντοπιστεί όμως και η διαφωνία με τις χώρες μέλη. Πώς θα προχωρήσουν αυτές. Προτείνει η συγγήτρια ένα όργανο συντονισμού με κάποια παραλλαγή θα πρέπει αυτό να γίνει δεχτό. Δεύτερο, δεν ξέρω αν έχει σχετικά σχέδια η Κομισιόν, αλλά θα είναι πάντως δύσκολο, γιατί τέτοιου είδους θεσμικά όργανα υπάρχουν στις χώρες μέλη και με περιφερειακές δραστηριότητες. Και καμιά φορά διαπιστώνονται εκεί και εγωισμοί, ιδίως δε για το διάστημα Διαπιστώνεται αυτό και στην Κομισιόν, δηλαδή υπάρχουν συναρμόδιες γενικές διευθύνσεις, όχι μόνο ο Γαλιλαίος αλλά και αλλού, που χρειάζονται σαφή συντονισμό και που δεν υπάρχει πάντα. Για τα έργα η κυρία Νίπλερ λέει για τον Γαλιλαίο και τον Κοπέρνικο, καθώς επίσης και για την παρακολούθηση των αποβλήτων στο διάστημα. Το ερώτημα τι θα κάνουμε με αυτά τα απόβλητα στο διάστημα Καλές είναι οι προτάσεις αυτές, αλλά και δαπανηρές. Πρέπει ωστόσο ταυτόχρονα να προστατευτεί το διάστημα. Εκεί πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Κατά τα λοιπά, αναμένω με ενδιαφέρον τη συζήτηση με τους και τις συναδέλφους. Ελπίζω ο Γαλλέος έτσι να μπορέσει να προχωρήσει, διότι διαπιστώνω ότι Κίνα και Ρωσία, παρόλο που πέσανε τρεις ρωσικοί δορυφόροι, δεν κοιμούνται και αρπάζουν κάθε ευκαιρία για να προχωρήσουν. Ευχαριστώ. Τζόνσον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Και ευχαριστώ ε, και τον κύριο Έλλερ που μας παρουσίασε την πρόταση ηγετρίας. Είναι πολύ καλό σημείο εφετηρίας για τη διαστημική βιομηχανία. Έχω κάποιες ε, συμπληρωματικές ερωτήσεις και κάποια σχόλια. Ο κλάδος αυτός είναι ιδιαίτερα καινοτόμος και μάλιστα ε, διασπέρει τεχνολογία και σε άλλους σημαντικούς τομείς. Το διάστημα θα δώσει μεγάλη όθηση και η διαστημική βιομηχανία σε πολλούς κλάδους της βιομηχανικής δραστηριότητας. Η διαστημική βιομηχανία βρίσκεται στο προπύργιο της ε, καινοτομίας και γι' αυτό και θα πρέπει να του δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και στα πλαίσια της ε, προσπάθειάς μας ε, για οικονομική ανάκαμψη και για τόνωση της απασχόλησης. Έχουμε πολλές προκλήσεις. Θα πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ της διαστημικής έρευνας και της ανάπτυξης των προϊόντων, ώστε να έχουμε αποτελεσματική θέση εμπειρία και καλή συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημιακών και των βιομηχάνων. Η κατάσταση βέβαια διαφέρει από χώρα σε χώρα Άλλωστε πρόκειται για ένα τομέα που κυριαρχείται από λίγες πολυεθνικές και από πολύ μεγάλους ομίλους, θα πρέπει να υποστηρίξουν περισσότερο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να ενταχθούν και αυτές στην καινοτομία που είναι σημαντική για τη διαστημική βιομηχανία. Προσβλέπω στενή συνεργασία με την εισηγήτρια και ενστερνίζομαι την άποψη ότι η πρόταση του Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι πολύ φιλόδοξη, ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε καλύτερα με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ, κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε εδώ μια κατάσταση στην οποία η Ευρώπη έχει μια βιομηχανία και ένα κλάδο με υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Θα πρέπει λοιπόν πάση θυσία να διατηρήσουμε αυτή την ευρωπαϊκή υπεροχή, ε, πρικοδοτώντας τον κλάδο με τους απαραίτητους πόρους για να ανταπεξέλθει στην αποστολή του και στους στόχους του. Θα ήθελα να επισημάνω κάποια θέματα έρευνας που είναι σημαντικά για το μέλλον και θα πρέπει να προωθηθούν. Καταρχήν, ε, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο πολύ σημαντικό θέμα, όπως και η ασφάλεια των δεδομένων που ανταλλάσσουμε σήμερα μέσω των δορυφόρων πλοήγησης. Θα πρέπει αυτές τις επικοινωνίες να τις στεγανοποιήσουμε απέναντι σε παρεμβολές ή παρακολούθησης που θα μπορούσαν να έχουν πολύ αρνητικές συνέπειες. Έχουμε και το θέμα της ε, δορυφορικής ε, παρακολούθησης ε, του satellite tracking. Πολύ σημαντικό θέμα εδώ είναι η συνειδητοποίηση ότι υπάρχει μεγάλη εξάρτηση σε θέματα διαστημικής τεχνολογίας. Οπότε θα πρέπει να φροντίσουμε για την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια αυτών των θεμάτων. Και θα ήθελα να αφαιρθώ και σε μερικά άλλα θέματα. Θέλουμε εξειδικευμένη έρευνα προκειμένου να μειωθούν τα διαστημικά απόβλητα. Έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρξει ένα σημείο ε, διασύνδεσης έτσι ώστε να μπορεί να γίνει εκτόξευση με βάση μία διεθνή συμφωνία, αλλά για μένα θα πρέπει να ε, μην βρίσκονται πλέον σε τροχιά είτε αυτοί οι δορυφόροι, ο κύκλος των οποίων έχει τελειώσει, είτε θράψματα αυτών. έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί και ε, το θέμα σύγκρουσης όταν προκύπτει. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε το θέμα μέσα σε ένα συγκεκριμένο ε, χρονισμό. Δηλαδή αυτό που έχει σημασία είναι οι ηλιακές αυτές θύελες, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν και πώς μπορεί να συνεχιστεί η έρευνα για τους εκτοξευτές με βάση τα ε, διαστημικά στοιχεία τα οποία μπορεί να διαθέτουν και μη Underdaughter. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που λαμβάνω και εγώ μέρος στη συζήτηση, γιατί αφορά την ε, μελλοντική και αποτελεσματική διαστημική βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την ε, καθοδήγηση της κυρίας Σνίμπλερ. Πολύ σημαντικός κλάδος με μεγάλα πλονεκτήματα ε, όχι μόνο για, τον, για την Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Κοινότητα, αλλά και για την παγκόσμια. Έχει και οικονομικά ωφέλη που τα ακούσαμε από τους συναδέλφους. Δημόσιες επενδύσεις αποτελούν από, την αρχή τη βάση της, του διαστημικού αυτού κλάδου και του ευρωπαϊκού, ιδιαίτερα για τις πιο ακριβές δραστηριότητες όπως είναι η εκτόξευση, η κατασκευή διαστημικών σκαφών, αεροσκαφών. Με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαράζουμε το δρόμο για μια ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική που θα αποφέρει και οικονομικούς και κοινωνικούς καρπούς. Πολύ σημαντική έκθεση κυρίας Νίμπλερ και από θέματα από άποψη πολιτικής και άποψη θεσμικού πλαισίου και προσβλέπω σε βάθηση της συζήτησης. Θέλουμε βέλτιστη χρήση των δεδομένων από την παρακολούθηση της γης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει για τα διαστημικά θράψματα να δίνονται σχεδόν δωρεάν ή δωρεάν οι πληροφορίες και πιστεύω ότι είναι σημαντικό αυτό γιατί ούτω ή άλλω με δημόσιου φόρου γίνεται η έρευνα. Οπότε είναι λογικό το κοινό να έχει δωρεάν πρόσβαση σε αυτά. Σε ό,τι αφορά το Διαστημικό Ταμείο, η ανάπτυξη του διαστημικού τουρισμού είναι ένα πολύ ε, ενδιαφέρον θέμα και το πρόγραμμα Μόρις ε, ε, είναι αποσπά ιδιαίτερα την προσοχή και μάλιστα ήδη την περασμένη εβδομάδα έχουμε ξεκινήσει στο ειδικό Υπουργείο μία πρόκληση για υποβολή ενδιαφέροντος. Ποιοι θέλουν να επωφεληθούν από τέτοιο διαστημικό τουρισμό. Θα πρέπει όμω όταν αναπτύξουμε αυτά τα διαστημικά προγράμματα να έχουμε υπόψη το κοινό συμφέρον, να μην επωφεληθούν μόνο λίγοι επιλεκτοί πολιτικοί κάποιοι δισεκατομμυρίουχοι. Επίση, θα πρέπει να περιλάβουμε πολύ περισσότερε επιχειρήσει και κυρίω μικρομεσαίε επιχειρήσει. Να εξετάσουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία ότι στο, ευρωπαϊκό έδαφο να έχουμε μια βιώσιμη διαστημική βιομηχανία που θα στηρίζεται σε μεγάλη προσφορά και σε δυναμική ζήτηση. Σε ό,τι αφορά την κατανομή του φάσματος, και της ε, ασφαλής ε, συχνότητε για διαστημικές επικοινωνίες, ε, εξασφαλίζοντας φυσικά τη διαφοροποίηση. Είναι σημαντικά βέβαια οι στρατηγικοί φορείς μονοπολούν σχεδόν αυτά τα θέματα, ενώ θέλουμε και μη στρατηγική χρήση. Έχουμε δυστυχώς σπάνι του τις συχνότητες. Γι' αυτό και θα πρέπει να αναπτύξουμε και άλλες τεχνολογίες όπως είναι οπτικές σύνες και άλλες. Σας ευχαριστώ και περιμένω περαιτέρω συνεργασία. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω εν συντομία ότι ευχαριστώ ιδιαίτερο στην εισηγήτρια για την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσής της και ευχαριστώ επίσης θερμά όσοι έλαβαν το λόγο γιατί εξέφρασαν ενθουσιώδη σχόλια σε μεγάλο βαθμό για την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με τα σχόλιά σας και με τα βασικά σημεία της έκθεσης. Πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο θέμα του συντονισμού. Ένα ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Νοέμβριο του 2012 μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μία ανακοίνωση που ακριβώς αφορά τις σχέσεις ε, της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ώστε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τους διαθέσιμους πόρους που θα είναι περισσότερο στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλίσουμε σχέσεις ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και των κρατών μελών που θα είναι πιο στενές, πιο έντονες και θα εξασφαλίσουν την βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ε, για θέματα διαστήματος. Ευχαριστώ. Ich möchte nur Επιθυμώ μόνο να ευχαριστήσω όλες και όλους εξ ονόματος της κυρίας Νίπλερ. Έχουμε κάνει τη συζήτηση για το πρόγραμμα έρευνας με πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις, ωστόσο συμφωνήσαμε εν τέλει και είπαμε ότι για την διάθεση των κονδυλίων ένα μέγα θέμα είναι ο συντονισμός και τελικώς και το Συμβούλιο μετά από πολλές συζητήσεις το δέχθηκε. Ωραία. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Έλλερ. Υπενθυμίζω ότι η προθεσμία υποβολή τροπολογιών είναι Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Περνάμε στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης, αλλαγή του κανονισμού 912 κάθετος 2010 ε, για τη σύσταση οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS. Η έκθεση αυτή ότι πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές απεστάλλει για μετάφραση 17 Ιουλίου. Σήμερα έχουμε για πρώτη φορά την ευκαιρία να συζητήσουμε το περιεχόμενο. Η υποβολή τροπολογιών. Η προθεσμία είναι η 19η Σεπτεμβρίου και θα ψηφίσουμε στις 14 Οκτωβρίου στην Επιτροπή. Με τους σκιώδεις έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και μας επέτρεψε να προχωρήσουμε την εργασία μας χωρίς να υπάρξουν προστριβές σε τεχνικό επίπεδο στις 26 Ιουνίου συναντηθήκαμε και για να έχουμε μία πρώτη ανεπίσημη ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων με την Επιτροπή. Ο οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS θα θυμόσαστε ότι δημιουργήθηκε το 2004 και βρίσκεται στην Πράγα στη νέα του έδρα από την 1η Σεπτεμβρίου του 2012. Πρωταρχική στόχη είναι η εγγύηση του Ευρωπαϊκού Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης, προωθώντας τα δημόσια συμφέροντα επαρκώς και η χρηματοδότηση να χρησιμοποιηθεί σωστά. Ο κανονισμός που εγκρίθηκε το 2008 ανέθεσε στον οργανισμό την ε, διαπίστευση συστημάτων ασφαλείας. Τώρα που ο οργανισμός θα λειτουργήσει πλήρως και που το πρόγραμμα Γαλιλαίος θα τεθεί πλήρως σε εφαρμογή, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την αυτονομία και των δύο οργανισμών. Η πρώτη επιτροπή στοχεύει στο να ορίσουμε καλύτερα τη διάρθρωση του οργανισμού και την ευθύνη των εσωτερικών οργάνων. Πέρα από την ευθυγράμμιση του κανονισμού με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι 44 τροπολογίες για την βελτίωση και τον καλύτερο ορισμό της δραστηριότητας και της διαδικασίας ευθύνης και ελέγχου στα πλαίσια του οργανισμού. Υπάρχουν έξι σημεία που θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους και μία σειρά τροπολογιών που στοχεύουν στην ευθυγράμμιση του κειμένου του κανονισμού με την κοινή προσέγγιση των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τη στιγμή έγκρισης της ε, πρότασης βρίσκονται στη διαδικασία ε, ε, γνωμοδότησης και τελικής έγκρισης επειδή δεν θέλουμε να υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων, πολλές τροπολογίες ορίζουν καλύτερα αυτή την πλαισίωση. Προβλέπεται ένα άρθρο ad hoc το 22α που περιλαμβάνει και διάφορες συστάσεις που εμπεριέχονται στην ε, ε, έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου του 2012. Θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός ε, ρόλων μεταξύ εκτελεστικού διευθυντή και ε, προέδρου της διαδικασίας διαπίστευσης και ασφάλειας. Επίσης υπάρχουν ειδικά άρθρα για τους απεσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες καθώς και το προσωπικό γενικότερα. Ενισχύεται η διαφάνεια έτσι ώστε ετήσια και πολυετή προγράμματα δραστηριότητας να περιέχονται καθώς και εσωτερικοί κανονισμοί οι οποίοι δημοσιοποιούνται. Τέλος, πολλές τροπολογίες ενισχύουν τη διαδικασία ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το, ρόλο του Γενικού Διευθυντή και του Προέδρου θεμάτων ασφάλειας. Επίσης προβλέπονται διορθωτικά μέτρα έτσι ώστε το, σύστημα, το κείμενο συγγνώμη, είναι συμβατό με άλλα συστήματα και οργανισμούς. Ο κ. Γκλάντε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω και ε, τίποτε σπουδαίε παρατηρήσεις. Καλά συνεργαστήκαμε. Δύο ερωτήσει μόνο σχετικά με τροπολογίες δικέ σα στην τροπολογία σας 31 για θέματα κανονισμού και πιστοποίησης ασφάλειας. Εμένα μου αρέσει η διαφάνεια. Μήπως εδώ όμως η υπερβολική διαφάνεια μπορεί να βλάψει. Γι' αυτό ρωτώ. Γιατί λέτε ότι πρέπει να δημοσιεύεται ο κανονισμός. Αυτό αναφέρεται μόνο σε αυτό ή προτίθεστε να ζητήσετε δημοσίευση και άλλων πραγμάτων. Επίσης, στην σύγκρουση συμφερόντων, στην υπαριθμόν 4, τα αναπτύσσετε υπερβολικά, ώστε μου προκαλείτε την ερώτηση υπήρξαν προβλήματα σχετικά σε κάποιους οργανισμούς και γι' αυτό αυτό είναι ένα είδος αντίδρασή σας. Αυτές τις δύο ερωτήσεις έχω. Κατά τα άλλα είμαι σύμφωνος η Πρόεδρος. κυρία Χολ, ευχαριστώ. είμαι και εγώ σύντομη. Χαιρετίζω την έκθεσή σας. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε πλήρη διαχωρισμό μεταξύ των διαφόρων πτυχών του GNSA και ε, της αρχής που εκδίδει τις ε, άδειες ασφάλειας. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι θέλουμε να αποκαταστήσουμε πλήρως ε, ένα απόλυτο διαχωρισμό. Η μόνιμη επιφύλαξη αφορά την διατύπωση ιδιαίτερα της τροπολογίας σας γιατί είναι αρκετά βαρύγδοπη διατύπωση και διαρωτάμε αν θα μπορούσαμε να επανέλθουμε σε αυτό που συμφωνήσαμε για την Ενίσα. Γιατί καταλήξαμε σε ένα σε ένα κείμενο που καλύπτει το θέμα της ε, σύγκρουσης συμφερόντος και στα πλαίσια του οργανισμού Ενίσα. Μήπως λοιπόν ε, θα πρέπει να ευθυγραμμιστούμε με τα όσα είχαμε αποφασίσει εκεί. Είναι σημαντικό και θεωρώ σωστό που εφαρμόζουμε τις συστάσεις ε, για τα, την εναρμόνιση ό,τι αφορά τους οργανισμούς και τη χρη, χρησιμοποίηση των βέλτιστων πρακτικών σε ό,τι αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Γιατί έχουμε πολλούς οικονομικούς οργανισμούς και μάλιστα είχαμε ε, συνεντεύξει στο Κοινοβούλιο και ακροάσει με του διοικητέ ε, ε, αυτών των οργανισμών στο Κοινοβούλιο, θα θέλαμε αντίστοιχη ακρόαση να διοργανωθεί και στην περίπτωση αυτή. Επίσης, ε, στηρίζω την πρότασή σας ότι το σώμα αυτό ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός θα πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα σε ό,τι αφορά την ίση συμμετοχή των δύο φύλων, η ισόρροπη εκπροσώπηση. Νομίζω ότι είναι πολύ ορθολογικό στόχος, σε καμία περίπτωση υπερβολικός και σας υποστηρίζουμε πλήρως. Η Επιτροπή θα ήθελε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς εσάς προσωπικά κυρία Πρόεδρε που δεχτήκατε να επεξεργαστείτε τη σημαντική αυτή πρόταση και έχετε εκφράσει την επιθυμία να συμφωνήσετε με το Συμβούλιο. Η έκθεση που υποβάλατε για μας αποτελεί καλή βάση για συζήτηση με το Συμβούλιο και προβλέπει ενίσχυση της GSA. Πρέπει να τονιστεί και πάλι ότι η ενίσχυσή της αποτελεί και σημαντικό στοιχείο, καινοτόμο στοιχείο, του κανονισμού GNSS, όπως θα αρχίσει να ισχύει από αρχές Ιανουαρίου του 2014. Έτσι, όλα τα μέτρα που προτείνετε εσείς κυρία Πρόεδρε, καθώς και οι τροπολογίες και που οδηγούν στην ενίσχυση του οργανισμού αυτού, για μας είναι καλόδεκτα. Είπατε ήδη ότι το σχέδιο της Κομισιόν προσπαθεί να επιτύχει τρία πράγματα. Πρώτα, την ενίσχυση σε προσωπικό του GSA είπα ότι από την αρχή του Ιανουαρίου 2014 αρχίζει νέα φάση για τον οργανισμό και για τον Γαλλίο και τον Κοπέρνικο. Δεύτερος στόχος της πρότασης της Κομισιόν είναι να υπάρξει σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων για τη λειτουργία αφενός και για την πιστοποίηση ασφαλείας από την άλλη μεριά, εντός του οργανισμού. Τρίτο, επίσης σημαντικό, όπως εξηγήσατε και εσείς άλλωστε, η εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για την νομική θέση των διαφόρων ευρωπαϊκών οργανισμών. Επαναλαμβάνω ότι είναι καλόδεκτες οι προτάσεις σας. Για τις επιμέρους διατυπώσεις μπορεί κανείς ακόμη αν θέλετε να συζητήσει. Αλλά δεν είναι τόσο πολύ το θέμα αυτό. Τονίζω και πάλι ότι από 1η Ιανουαρίου 2014 η Γενική μας Διεύθυνση αναλαμβάνει την διαχείριση του έγνος και επομένως μέγα βάρος για την άνευ τριβών διαχείριση του συστήματος, ενός συστήματος από το οποίο θα εξαρτηθεί στο μέλλον ακόμη περισσότερο η ασφάλεια των αεροπορικών επικοινωνιών. Δεύτερον, για το Γαλιλαίο που είναι πιο μακροπρόθεσμο σχέδιο, ο στόχος είναι το 2017, αρχίζει όμως η Γενική Διεύθυνση ήδη από σήμερα να ασχολείται και εκεί θα είναι απαραίτητο να ενισχυθεί σε προσωπικό, σε στελέχωση η GSA. Ολοκληρώνω τώρα λέγοντας ότι η πρότασή σας μας βρίσκει σύμφωνο. ελπίζουμε να συμφωνήσουν και τα άλλα μέλη σας, έτσι ώστε το δυνατόν συντομότερο να μπορέσουμε να αρχίσουμε τη συζητήσει με το Συμβούλιο για την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ευχαριστούμε την ε, Επιτροπή σας. Υπενθυμίζω ότι η ημερομηνία υποβολής τροπολογιών είναι η 5η 19 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι σε σχέση με τη, τους παρεμβάσεις Γκλάντ και Χολ θα λάβω υπόψη τις ε, παρεμβάσεις σας στην ε, περαιτέρω επεξεργασία του θέματος. Όπως ε, κατανοείτε, θέλαμε να φτάσουμε σε ορισμένους στόχους. Ένας από αυτούς είναι και η διαφάνεια. Τροπολογία 31 που σχετίζεται όχι μόνο με τον εσωτερικό κανονισμό, αλλά και την ετήσια έκθεση και το πρόγραμμα εργασίας που αποτελούν δημόσια έγγραφα. Η τροπολογία 4 σχετίζεται με την ετήσια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Αλλά βεβαίως πρόκειται για δύσβατα έγγραφα και γι' αυτό πιστεύω ότι με τροπολογίες θα δούμε πώς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους διαφάνειας, κυρίως με ε, βάση τα συναφή έγγραφα και κανονισμούς που έχουν μέχρι τούδε εγκριθεί έτσι ώστε το κείμενο να είναι απόλυτα σαφές με τη συνεργασία σας. μέσα στα πλαίσια της ε, κοινή αυτής ε, διαδικασίας και διεργασιών. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Περνάμε τώρα στην έκθεση Τόγια, η οποία αντικαθίσταται από το συνάδελφο Πρόντι σε σχέση με την ασφάλεια καταναλωτικών προϊόντων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το πακέτο για την ασφάλεια προϊόντων που εγκρίθηκε στις 13 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους θέτει ως στόχο μία νέα νομοθετική τάξη έτσι ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν σωστά, να εφαρμοστεί σωστά το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων και για την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς. Ο βασικός στόχος της ε, πρώτας Επιτροπής είναι να διασφαλίσει την θέση στην αγορά μόνο ασφαλών προϊόντων χωρίς να υπάρχει κατακαιρματισμός της αγοράς και αρνητική επιρροή ε, διαφόρων ε, προδιαγραφών. Το κείμενο θα ληφθεί υπόψη διεξοδικά και από την ΙΜΚΟ και από τις άλλες επιτροπές ε, ΕΜΒΙ, ΙΝΤΑ, ΕΜΒΙ και ΓΙΟΥΡΕ. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε μία ισορροπία σε σχέση με την ερμηνεία ε, των προϊόντων αυτών της ε, νομοθεσίας για τα προϊόντα αυτό χωρίς να, υπάρξουν, να υπάρξει διοικητικός ε, φόρτος. Η πρόταση αφορά τις γενικές προδιαγραφές ασφάλειας, σύνθεση, συσκευασία, χρήση και κινδύνους. Τη στιγμή που δεν υπάρχουν ειδικά νομοθετικά πλαίσια όπως ισχύουν για τα παιχνίδια, τα καλλιντικά, ε, τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και λοιπά. βάλουμε υπόψη και το δίκτυο διανομής έτσι ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες πληροφορίες ε, τις οποίες να γνωρίζει ο καταναλωτής. Σε σχέση τη γνωμοδότηση της Επιτροπής θεωρήθηκε σκόπιμο να σταθούμε σε ορισμένες ειδικέ πτυχές που σχετίζονται με την προστασία των καταναλωτών και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Θα ήθελα να τονίσω ορισμένα σημεία ο ορισμός του ευάλωτου καταναλωτή. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε μία πρόταση πρωτοβουλίας ε, τονίζοντας θέματα ασφαλείας ιδιαίτερα σε αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση, δηλαδή τους, ε, τους ευάλωτους καταναλωτές. Ως προς συνάδελφο λάβαμε υπόψη ε, τα παιχνίδια τα οποία είναι δελεαστικά, τα παιχνίδια που είναι δελεαστικά για τα παιδιά και τα οποία πολλούνται επιγραμμικά, τα οποία δεν είναι πάντα ασφαλή. Μας ενδιαφέρει υπόψη, το πώς θα λαμβάνει υπόψη η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για να υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια ασφάλεια για τους καταναλωτές και η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών έχει σημασία η ανιχνευσιμότητα και η προέλευση τροπολογίες 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 16 που επιτρέπουν την διασφάλιση της προέλευσης έτσι ώστε η παραγωγή να αναφέρουν επαρκή στοιχεία έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι για τις ποιοτικές προδιαγραφές. Θα πρέπει επίσης να, να τηρηθεί η αρχή της αμοιβαιότητας μεταξύ προϊόντων που παράγονται στην Ευρώπη και εισαγωμένων, για να μην υπάρχει διάκριση κατά ορισμένων επιχειρήσεων και υπάρξει δίκαιο εμπόριο παγκοσμίω. Ο κανονισμός θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί επιπρόσθετος διοικητικός φόρτος που θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις για να δημιουργηθούν κοινοπραξίες που θα λαμβάνουν υπόψη το εμπλεκόμενο ε, κόστος, τροπολογίες 1 και 5. Το κείμενο θα μπορέσει να βελτιωθεί με τροπολογίες και θα ήθελα να μου δώσουν, να μου υποδείξουν οι συνάδελφοι και νέες τροπολογίες. Ε, Κόρχολα. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Εγώ είχα ασχοληθεί πριν από τρία χρόνια με το θέμα αυτό της ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων. Είμαι και οδησηγήτρια ε, στην ΙΜΚΟ ε, για την έκθεση Αλντεμόζε που εξέταζε την αναθεώρηση της ε, οδηγίας για την γενική ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων. Οπότε κάποια στοιχεία αναμφίβολα θα τα επαναλάβουμε. Η νέα πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπάθησε να αντιμετωπίσει τις προηγούμενες αδυναμίες και τα παραθυράκια της προηγούμενης οδηγίας και να λάβει υπόψη κάποια σχόλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στάσεις από την έκθεση πρωτοβουλίας του. Βέβαια, έχω δύο επιφυλάξεις ως προς την έκθεση της εισηγητρίας και τον νέο κανονισμό σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική αναφορά της χώρας προέλευσης. Αυτή είναι η πρώτη επιφυλαξή μου. Έχει συζητηθεί το θέμα Πολάκης και είναι ένα ζήτημα πολιτικό που διχάζει τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του καταναλωτή και τη συνειδητοποίηση της κατάστασης, φυσικά θα ήταν ιδιότητας να γνωρίζει ο καταναλωτής την προέλευση των προϊόντων. Βέβαια, η χώρα προέλευσης δεν δίνει ενδείξεις για την ασφάλεια του προϊόντος και μάλιστα παραπλανεί τους ε, καταναλωτές να θεωρούν ότι όντως το, όλα τα τμήματα του προϊόντος ε, γίνονται στη χώρα προέλευση. Γιατί η χώρα προέλευση εξαρτάται από τον τελωνιακό κώδικο. Είναι χώρα δηλαδή όπου ε, γίνεται η μεταποίηση του τελευταίου συστατικού του προϊόντος. Οπότε όλα τα υπόλοιπα αισθητικά μπορεί να μεταποιούνται, να παράγονται σε πολλές διαφορετικές χώρες. Οι παρασκευαστές επίσης δίνουν ε, διάφορες πληροφορίες ε, ή έναν αριθμό σειράς προκειμένου να γίνει ε, να εξασφαλιστεί η χρηλασιμότητα της αλυσίδας παραγωγής αλλά η αναφορά επιπλέον και της χώρας προέλευσης δεν βελτιώνει την εκλασιμότητα ενός ε, προϊόντος που δεν είναι ασφαλές. Οπότε θεωρώ ότι η αναφορά της χώρας προέλευσης είναι θέμα ετικέτας περισσότερο, όχι θέμα ασφάλειας του προϊόντος. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα του ορισμού των προϊόντων που είναι ελκυστικά στα παιδιά. Ο προσδιορισμό των προϊόντων αυτών και η δημιουργία επιπλέον κριτηρίων ασφάλειας για αυτά τα προϊόντα που είναι δελαστικά για τα παιδιά συζητήθηκε επίσης πριν από μια τριετία όταν εξετάζαμε την έκθεση τη πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχει αλλοιωθεί αρκετά αυτή η έννοια και δεν ξέρω αν είναι εύκολο ο νομοθέτης να καθορίζει τι θα πει ελκυστικό προϊόν για τα παιδιά. Δηλαδή μια τοστιέρα είναι Mickey Mouse ή ένα κερί μοιάζει με φράουλα ή ένα, ε, μια συσκευασία σαμπουάν ε, έχει επίσης μια εικόνα από κινούμενο σχέδιο είναι πιο ελκυστική για τα παιδιά. Το θέμα αυτό χρήζει ιδιαίτερη προσοχή ε, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, όπως προβλέπει το άρθρο 6.1. Βέβαια, είναι αξιέπαινη προσπάθεια και επιθυμία να εξασφαλίσουμε ε, τα προϊόντα για τα παιδιά. Αλλά αν ένα παιδί είναι πολύ μικρό για να ε, εξετάσει πώς χρησιμοποιείται μια τοστιέρα, περισσότερο είναι ευθύνη του γονέα να την ε, φυλάξει σε ασφαλές μέρον παρά να επιβάλλουμε ιδιαίτερη, ιδιαίτερα κριτήρια ασφάλειας για την επικίνδυνοτητα τέτοιων προϊόντων. Πάντως χαιρετίζω την πρόθεση αυτή που βελτιώνει κατά πολύ την κατακαιρματισμένη σημερινή νομοθεσία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την κυρία Τόγια για την έκθεσή της για το σχέδιο το οποίο μας παρουσίασε δηλαδή ο κύριος Πρόντι. και οι δύο, τροπολο... Ε, αρμόδιες επιτροπές ε, θα καταθέσουν παρόμοιες τροπολογίες γιατί όλοι συμφωνούμε ότι η πλέον γραφειοκρατία βλάπτει την οικονομία και φυσικά παρεμποδίζει και την υλοποίηση του στόχου της ε, νομοθετικής αυτής ρύθμισης. Θέλουμε καλύτερη επιτήρηση των αγορών σίγουρα και ενισχυμένη ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, αλλά όχι περαιτέρω γραφειοκρατία. Τώρα να σχολιάσω τις τρεις προτάσεις της σου. Καταρχήν, τα προϊόντα που είναι δελαστικά για τα παιδιά. Ε, είναι αρκετά διασταλτική η ερμηνεία αυτού του προϊόντος. Μία, μία πολύχρωμη συσκευασία είναι αρκετή για να χαρακτηριστεί ένα προϊόντο ελκυστικό για τα παιδιά. Αμφιβάλλω. Νομίζω ότι ένα μεγάλο τμήμα τη ευθύνη το φέρουν οι γονεί. Δεν μπορούμε εμεί να υποκαταστήσουμε την ευθύνη των γονιών για επιτήρηση των παιδιών του και φύλαξη των προϊόντων. Σε ό,τι αφορά την αναφορά χώρας προέλευσης, είναι αρκετά επίμαχο αυτό το θέμα. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι ο στόχος του συγκεκριμένου κανονισμού δεν είναι η εμπορική πολιτική, αλλά η επιδίωξη της ασφάλειας των προϊόντων. Στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπονται κάποιες υποχρεώσεις των παραγωγών και των εισαγωγέων. Αν όμως δεν έχουμε ε, αξιολογήσεις ε, της εφαρμογής του κανονισμού θα δημιουργήσει μια επιπλέον τέτοια υποχρέωση, υπερβολικό άχθος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί μην ξεχνάτε ότι οι αποδέκτες αυτού του κανονισμού θα είναι μόνο μεγάλες ε, εταιρείες, αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ακόμη και αν μεγάλα τμήματα του προϊόντος παράγονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μπορούν να αναφέρουν ως χώρα προέλευσης ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τον Τελωνιακό Κώδικα. δεν μπορεί να ξέρει κανείς από πού προέρχεται η κάθε πρώτη ύλη του προϊόντος. Και η αναφορά της χώρας προέλευσης καλύπτει μόνο την τελευταία φάση της διαδικασίας παραγωγής, της διαδικασίας μεταποίησης. Οπότε δεν δίνει και πολλά στοιχεία ε, η πληροφορία της χώρας προέλευσης. Γι' αυτό και έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις για το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά τις προειδοποιήσεις ή το όριο ηλικία, για παράδειγμα, καλή η πρόθεση στη θεωρία, αλλά στην πράξη θα δημιουργήσει προβλήματα και έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Γιατί δεν αναφέρεται για κάθε ομάδα προϊόντων τι προειδοποίησεις χρειάζονται. Νομίζω ότι ήταν καλύτερη εδώ και προτιμότερη η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εδω και προτιμοτερη η προταση ευρωπαικης επιτροπης οπως το άρθρο 6 μιλά με καλύτερο τρόπο για την κάλυψη αυτών των προειδοποίησεων. Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε ομόφωνη λύση για τα προβλήματα αυτά και ευχαριστώ την εισηγήτρια για την αξιέπαινη προσπάθειά της. Ευχαριστώ επίσης θερμά και τους σκιώδης εισηγητές. Η κυρία Άντερ Και εμένα με απασχολεί το θέμα της ε, ασφάλειας των ε, καταναλωτικών προϊόντων άκουσα ότι λιγότεροι Σουηδοί αρρωσταίνουν ε, λόγω της ε, κατανάλωσης τροφίμων αλλά την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι έχουν ε, βελτιωθεί οι προδιαγραφές ασφαλείας. Αλλά υπάρχουν ορισμένα σημεία που θα ήθελα να θίξω. Συμφωνώ απόλυτα με τα θέματα που ε, οι συνάδελφοι φιλελεύθεροι και ο συνάδελφος του ΕΛΚ σε σχέση με την αναγνώριση προέλευσης. Ίσως είναι θέμα σήμανσης, αλλά όχι θέμα ασφάλειας και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Επίσης με εκπλήσει το πώς ορίζει η Επιτροπή την ανείχνευση των προϊόντων που δεν είναι ασφαλή θα πρέπει να ξέρουμε ποια προϊόντα είναι ασφαλή, αλλά τα ε, μη ασφαλή ε, είτε ανοιχνεύονται είτε όχι υπάρχουν. Θα ήθελα να ε, αλλάξει η διατύπωση του κειμένου. Μιλήσαμε για απολύσεις από δεύτερο χέρι και αυτό με απασχολεί κάπως διότι το έθιξε και ο κύριος Κρόιτσμαν. Σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχουν έψιλων ή πολίτες που πολλούν προϊόντα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει κατάλληλη πιστοποίηση και ίσως εάν υπάρξει φόρτος δεν προβούν σε αυτές τις πωλήσει. Νομίζω ότι οι πωλήσει ε, από δεύτερο χέρι θα πρέπει να προωθούνται πάντα και να μην αναχαιτίζονται. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς οι πωλήσει ε, ε, από δεύτερο χέρι που είναι νόμιμες μπορούν να ε, έχουν ένα ευρύτερο πλαίσιο μέσα στα πλαίσια αυτής της δραστηριοποίησης, δηλαδή η Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για τα σχόλια. Χαιρόμαστε για τη συζήτηση που γίνεται σήμερα. Θα ήθελα να πω ότι τα θέματα που εθίγησαν σήμερα είναι τα ίδια με αυτά που αναγνωρίζουν τα κράτη-μέλη. Ως προς την έκθεση καθεαυτή χαιρόμαστε διότι γίνονται προσπάθειες βελτίωσης της πρότασής μας όταν μιλάμε για τον ορισμό του ευάλωτου καταναλωτή ή την αναφορά ε, προϊόντων που είναι τελεαστικά προς ε, τα παιδιά. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί διότι το Κοινοβούλιο μας επέσυρε την προσοχή σε αυτό το θέμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οδηγία του 2005 για τις αθέμητες πρακτικές καλύπτει αυτό το ζήτημα και πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να ορίσουμε το, την έννοια του ευάλωτου καταναλωτή. Ε, διενεργείται μία μελέτη και αναμένουμε τα αποτελέσματα του 2014. Αυτό είναι ευαίσθητο θέμα. Το ίδιο αφορά και τα προϊόντα που είναι δελεαστικά για τα παιδιά. Θα πρέπει να βελτιωθεί το κείμενο. Ως προς τη σήμανση περιπροέλευσης, το θέμα αυτό έχει συζητηθεί Πλιστάκης και θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίστηκε στην ε, πείρα της από το σύστημα έγκαιρης ε, προειδοποίησης γιατί και στον τομέα μη τροφίμων πάλι είμαστε επικεφαλής ενός συστήματος μέσα στα πλαίσια της έγκαιρης προειδοποίησης και ένα 10% των προϊόντων δεν την χάνει αυτή της διασφάλισης προέλευσης. 10% ε, είναι υψηλό ποσοστό. Όταν μιλήσαμε για την σήμανση προέλευσης, στην πρότασή μας λάβαμε υπόψη τη βελτίωση του συστήματος ανιχνευσιμότητας προϊόντων που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή αγορά. Μαθαίνουμε με βάση την πείρα μας. Τώρα ως προς την πρακτική και το εμπόριο θα ήθελα να πω ότι η σήμανση προέλευσης δεν αποτελεί κάτι το καινοτόμο, αποτελεί προαπαιτούμενο στην νομοθεσία των ΙΠΑ, Ιαπωνίας κλπ. Δεν είναι κάτι που ξεκίνησε στην Ευρώπη οι Ευρωπαίοι παραγωγοί πρέπει να τηρούν αυτές τις προδιαγραφές όταν ε, προβαίνουν σε εξαγωγές. Και αυτό για να απαντήσω σε ορισμένα από τα σημεία που θίξατε ως προς τις τροπολογίες ε, για την προέλευση των συστατικών θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ε, πείρα μας σε άλλους τομείς, στον τομέα των τροφίμων και ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο. Οι τρέχουσες πρακτικές βασίζονται στο βαθμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε ένα καθολικό σύστημα για την προέλευση και τη σήμανσή της. Γι' αυτό και η βασική πρόταση είχε περιοριστεί στο τελικό προϊόν όπου γίνονται και οι τελευταίες ουσιώδες ε, μεταβολές επί του προϊόντος. Ελπίζω αυτά τα στοιχεία να σας βοηθήσουν Είμαστε στη διάθεσή σας. Τέλος, σας ευχαριστούμε διότι το αντιμετωπίσατε αυτό το θέμα κατεπηγόντως για να λυθεί σε αυτή τη θητεία, για να μην χάσουμε τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο στην ε, εξασφάλιση ε, της ασφάλειας αυτής, της γενικότερης ασφάλειας των προϊόντων πρώτη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Δεν ε, θέλω να κρίνω θα αναφέρω αυτά τα στοιχεία στη συνάδελφο, διότι εκείνη γνωρίζει το θέμα εις βάθος, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι υποδείξεις. Ευχαριστούμε, υπενθυμίζω ότι την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι το πρόγραμμα υποστήριξης για διαμητήρηση και παρακολούθηση του διαστήματος η Αμέλεια Ντότερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που είμαι η συγγήτρια της πρότασης αυτής τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σύσταση ενός προγράμματο επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος. Ελπίζουμε ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα θα συμβάλλει στην ασφάλεια των αντικειμένων σε τροχιά και θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί και αλλού. Μάλιστα έχουμε ε, σημαντική θέση στην ε, εκτόξευση και ε, των δορυφόρων και θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτή τη δραστηριότητα, ιδιαίτερα να έχουμε το Γαλλαίο και το Κοπέρνικο, γιατί υπάρχει κίνδυνος θραυσμάτων ή τεχνικών αντικειμένων να συγκρουστούν με τους δορυφόρους μας. Τέτοιος κίνδυνος θα πρέπει να προσοβηθεί. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, η Επιτροπή και το Συμβούλιο και εγώ συγκεκριά συμφωνούμε με τα σχόλια αυτά και ελπίζω να έχετε λάβει και το έγγραφο εργασία. Όπω αναφέρεται εκεί, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση στερείται μια τέτοια υπηρεσία για την παρακολούθηση διαστημικών αντικειμένων και απειλείται με συμφόρηση. Απειλούνται με συμφόρηση πολλέ ορισμένε τροχέ. Έχουμε 70 εκατομμύρια ευρώ προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την χρηματοδότηση αυτού του προγράμματο. Οι φορεί τη βιομηχανία μα λένε ότι η έλλειψη κονδυλίων ίσω δημιουργήσει ε, αντικίνητρα για τις υποδομές, ενώ χρειαζόμαστε πολύ σημαντικές υποδομές όπως είναι αισθητήρε ε, ε, και δορυφόροι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν μία πλήρη ικανότητα SST ύψους 200 εκατομμύριων ευρώ, που είναι πολύ ψηλότερα από τα 70 εκατομμύρια που μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το δικό μας σύστημα παρακολούθησης και επιτήρησης. Άλλωστε και η Οικονομική και η Κοινωνική Επιτροπή ζήτησαν επιπλέον κονδύλια για τις επενδύσεις στις υποδομές ενός τέτοιου συστήματος, αλλά δεδομένου στις οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουμε και τις κρίσεις, όπως φαίνεται και από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις σχετικές συζητήσεις, και εξαιτία ε, των κριτηρίων ασφάλειας και ποιότητας ε, των δεδομένων, εγώ θα ήμουν έτοιμη να, ε, να υποστηρίξω την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έναρξη με τη δικτύωση των σημαντικών των διαθέσιμων πόρων και να την αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού. Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, θα πρέπει να δούμε πού, από πού θα εξασφαλίσουμε αυτά τα 70 εκατομμύρια ευρώ. Αν προσθέσουμε επιπλέον στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο μια νέα δημοσιονομική γραμμή, ίσω δημιουργηθούν προβλήματα. Ίσως θα πρέπει να, δούμε, να προσπαθήσουμε να βρούμε αυτά τα κονδύλια από το υπάρχον πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Το Γαλιλαίο είναι σημαντικό συνεισφορέα, όπω λέει και στο παράρτημα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ίσω και η στρατηγική για την ασφάλεια. Σε ό,τι αφορά το Κοπέρνικο. Θα είναι σημαντική συνεισφορά του στο SST, αλλά θα πρέπει να δούμε αν συμφωνεί το Συμβούλιο με προέλευση του κονδυλίου από εκεί. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένο σαφή προπολογισμό με πόρους που θα καλύπτουν όλα τα σκέλη της πρότασης και άλλα προγράμματα που ε, θα ε, χρειαστούν για το SST θα πρέπει να δούμε πώς θα συμβάλλουν στο όλο σύστημα. Επίσης μπορούμε να έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία με τους συναδέλφους της Επιτροπής Προϋπολογισμών και ιδιαίτερα την κυρία Καρβάλιο που είναι η συγγήτρια της γνωμοδότησης για το SST, το σύστημα δηλαδή παρακολούθησης και επιτήρησης ε, της κατάστασης στο διάστημα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν όσο καλύτερη αξιοποίηση των ικανοτήτων των κρατών μελών και σε ό,τι αφορά το τεχνικό επίπεδο. Στο άρθρο 3, τι ικανότητες θα χρησιμοποιηθεί. Καταρχήν υπάρχοντες ε, αισθητήρε όπως το γαλλικό και το γερμανικό σύστημα. Επίσης θα πρέπει οι τηλεσκόπια και δορυφόροι που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης ε, να μπορέσουν σε μεταγενέστερο επίπεδο να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα αν πληρούν τα τεχνικά κριτήρια και τα κριτήρια επιλογής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης θέλουμε να κλείσουμε την πόρτα για ε, ικανότητες και στοιχεία που θα μας χρειαστούν στο μέλλον. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στην απόφαση. Σε ό,τι αφορά τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα SST, ελπίζω να το συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους συναδέλφους ε, τι πληροφορίες, τι επιπλέον λεπτομέρειες θα πρέπει να προσθέσουμε στο κείμενο, ώστε να καλωθορίσουμε καλύτερα το, το πλαίσιο των μελλοντικών δράσεων. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό διαστημικών αντικειμένων, θα προτιμούσα δωρεάν με βάση το σύστημα Two Line Elements των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Επίσης θα ήθελα με τους συναδέλφους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητήσουμε τη δομή μιας υπηρεσίας SST. Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική πτυχή των δεδομένων θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ακεραιότητα και την ασφάλειά τους πώς θα βρει ισορροπία μεταξύ της μη ε, κοινοποίηση εμπιστευτικών στοιχείων αλλά και της ε, ανταλλαγής δεδομένων με ενδιαφερόμενους φορείς. Επίσης θα πρέπει να έχουμε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να βελτιώσουμε τις ε, υπηρεσίες. Και θα μπορούσαμε να έχουμε συνεργασία ε, με, και με ιδιωτικούς φορείς όπως την την Ένωση Στοιχείων Διαστήματος που περιέχει βάση δεδομένων με πολύ σημαντικές πληροφορίες από αισθητήρε και δορυφόρους. Αυτά και περιμένω τα σχόλια των συναδέλφων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Πρόντι έχει το λόγο. Ευχαριστώ για αυτή την ε, έκθεση ιδεών. Συμφωνώ απόλυτα με το κείμενο αυτό. Γιατί το διάστημα αποτελεί μία βασική πηγή αντιμετώπισης ε, κινδύνων και υπάρχει η πιθανότητα να μην έχουμε τη δυνατότητα να εγγυηθούμε συγκεκριμένες ε, υπηρεσίες αυτό μπορεί να προκληθεί από ενδεχόμενες συγκρούσεις. Το θέμα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί τάχιστα, διότι διατρέχουμε τον κίνδυνο ε, μίας ε, μείωσης παροχής υπηρεσιών, διότι μπορεί να υπάρξει ε, ε, να υπάρξουν πολλές χιλιάδες θραύσματα που προκαλούνται από μία σύγκρουση. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να γνωρίζουμε πού βρίσκονται αυτά τα θράψματα, αυτά τα σωματίδια, για να υπάρχει η δυνατότητα να υπολογίσουμε την πιθανότητα σύγκρουσης. Όπως προανέφερα, νομίζω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τηλεσκόπια έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι για τα στοιχεία και να μπορέσουμε να ελέγξουμε αυτά τα αντικείμενα, και να ξέρουμε ποιες είναι οι πιθανότητες σύγκρουσης και πώς θα λάβει η χώρα μια τέτοια σύγκρουση για τους δορυφόρους δηλαδή που μπορούν να τηλεοδηγηθούν. να τηλεκατευθυνθούν. Επίσης, θα πρέπει να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για την, να βγουν από τροχιά αυτά τα αντικείμενα ισοματίδια, διότι μόνο έτσι μπορεί να επιληθεί το θέμα. Τζόνσον. Ευχαριστώ και ευχαριστώ ιδίως την κυρία Άντερ Στότερ για τα όσα εξήγησε. Συμφωνώ με τις απόψεις που εκφράζονται στο έγγραφο εργασίας. Νομίζω ότι η κυρία Άντερ εργάστηκε με πολύ θετικό τρόπο. Άλλωστε συνεργάστηκε καλά και με μένα και με άλλους και οδησίγητες. Θέλω να έρθω σε ένα θέμα που νομίζω δείχνει και τον επίγοντα χαρακτήρα όλης αυτής της συζητήσεως. Ένα θέμα πάντως που συζητήθηκε και πριν, ότι δηλαδή οι επιμέρους χώρες μέλη δεν μπορούν να αναλάβουν το βάρος τις προσπάθειες αυτής. Γι' αυτό χρειάζεται συνεργασία στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στο παγκόσμιο επίπεδο. Και γι' αυτό χρειάζεται να βρεθούν οι σωστοί τρόποι, οι σωστές φόρμουλες συνεργασίας. Να βρούμε τρόπους συνεργασίας ώστε να μπορέσουμε να έρθουμε στο ύψος της προκλήσεως. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια να διευκρινίσουμε την πορεία αυτή τρόπους λήψεως αποφάσεων, εμπιστευτικότητα των δεδομένων καθώς και χρηματοδότηση. Μπορούμε να κάνουμε καλή δουλειά στην βάση του εγγράφου που μας έχει υποβληθεί. Και εδώ νομίζω πρέπει να εμβαθύνουμε. Πάντως στο σύνολό της η πρόταση Στότερ είναι σωστή. Πολύ καλή δουλειά κύριε Στότερ. Ο κύριος Ρούμπικ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ με τη σειρά μου την κυρία Στότερ για αυτή την πρώτη έκθεσή της εκπροσωπώ την συναδελφό μου εδώ η οποία δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα. Η έκθεση είναι σημαντική για την βιομηχανία, είναι σημαντική ακόμη περισσότερο για την βιομηχανία του μέλλοντος, διότι ανοίγονται νέες επιχειρηματικές δυνατότητες, ιδίως στον τομέα των επικοινωνιών. Βλέπουμε πως έχουν εκτοξευθεί στα ύψη οι όγκοι των δεδομένων που μεταφέρονται με μεγάλη ταχύτητα, πόσο σημαντική είναι αυτή η όγκη, αυτά τα μεγέθη για την ανάπτυξη της οικονομίας. Μπορούν βεβαίω να προκληθούν και μεγάλες ζημίες. Στο διάστημα γίνονται λιγμοί που μπορούν να οδηγήσουν και σε ατυχήματα και επομένως σε σημαντική βλάβη υφισταμένων δομών. Πρέπει να έχουμε εικόνα ώστε να μπορούμε στο μέλλον να αντιδρούμε σωστά και ιδίως έγκαιρα. Ακόμα δεν έχουμε σε επαρκή βαθμό τις δομές αυτές. Γι' αυτό και νομίζω ότι απαιτείται διεθνή συνεργασία που αυτή πρέπει να λάβει την πρώτη προτεραιότητα. Με τα προγράμματα Γαλιλαίος και Κοπέρνικος καθώς και εμβληματικές πρωτοβουλίες είμαστε παρόντες στο διάστημα. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία αυτή και στο μέλλον να αναζητήσουμε τις ορθές απαντήσεις, ιδίως στις τηλεπικοινωνίες, όπου θα σημειωθεί ακόμη μεγάλη ανάπτυξη. Το ίδιο στον τομέα της πλοήγησης. Και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των δεδομένων, χρειάζεται να καταβληθούν νέες προσπάθειες. Ειδικά τους τελευταίους μήνες, αυτά που είδαμε από την άποψη της ηλεκτρονικής της ασφάλειας μάλλον της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι πολύ σημαντικά και εκεί πρέπει να οριστούν κιόλας οι τρόποι μεταφοράς των δεδομένων. Αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την περαιτέρω συζήτηση και νομίζω ότι ο τομέας αυτός θα είναι κρίσιμος για το μέλλον μας. Ευχαριστώ. Κυρία Καρβάλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αμέλη Ανταρστότηρ για την πολύ καλή έκθεση που μας υπέβαλε. Για το έγγραφο εργασία της που σε μεγάλο βαθμό αφηγραμμίζεται και με τη δική μου γνωμοδότηση που είμαι αρμόδια για την αντίστοιχη έκθεση το, για το SST στην Επιτροπή Προπολογισμών, αλλά και για την έκθεση για το Γαλιλαίο και το Κομπέρνικο. Και ευελπιστώ ότι χάρη και στη συνεργασία με τους κοιόδης ηγητές μας θα καταφέρουμε να βρούμε λύση στις δυσχερείς συνθήκες που διανύουμε, και όπως είπε και η Αμέλια Άγγελς Τότε, 70 εκατομμύρια δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά μπορούμε τουλάχιστον να χρηματοδοτήσουμε κάποιες προπαρασκευαστικές δράσεις. Προσβλέπω σε στενή συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών ώστε να εξασφαλίσουμε τον καλύτερο δυνατό προπολογισμό και να βρούμε φυσικά και τις πηγές χρηματοδότησης. Ευχαριστούμε Μαρία Καρβάλιο, ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και την εισηγήτρια για το πολύ καλό έγγραφο εργασία που μοίρασε. Θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα σημεία και να διευκρινίσω την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. νομίζω ότι αναφυσβήτητα έχετε συνειδητοποιήσει ότι η πρόταση αυτή, σε αντίθεση με την πρόταση για το Γαλιλαίο και τον Κοπέρνικο, δεν ζητά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την θέσπιση αυτής της υπηρεσίας. Απλώς θέλουμε ένα πρόγραμμα για να στηρίξουμε τις προσπάθειες των κρατών μελών με απότερο στόχο την ε, δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος SST, δηλαδή επιτήρηση και παρακολούθηση ε, της κατάστασης του διαστήματος. Είναι σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, γιατί αφορά την ε, δομή της πρότασης και το επίπεδο λεπτομεριών που μπορεί να παρουσιάζει. Γιατί μπορούμε να πούμε σε κράτη μέλη ότι αν συνεργαστείτε με τέτοιο τρόπο και για τέτοιο αποτέλεσμα θα μπορούσαμε να παράσχουμε αυτά τα κονδύλια. Η προσέγγιση αυτή ε, αλλάζει πολύ και το είδος των προτάσεων που μπορούμε να περιλάβουμε σε ένα τέτοιο έγγραφο. Ο προϋπολογισμός είναι περιορισμένος όπως είπατε και όλοι οι προλαλήσαντες επισήμαναν το σχετικά χαμηλό προϋπολογισμό και ευχαριστώ τους Ευρωβουλευτές για την υποστήριξή τους και την προθυμία τους να βρούμε λύση. Ο... Η συγκέντρια μας μίλησε για μια εμβριακή προσέγγιση. Είναι αρκετά δόκιμη αυτή η ορολογία. Το... Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αξιοποιήσουμε τη δικτύωση και την απαραίτητη συνεργασία για να δημιουργήσουμε στη συνέχεια το σύστημα. Χωρίς προηγούμενη δικτύωση ε, και ανάπτυξη των ικανοτήτων μας δεν θα καταλήξουμε ποτέ σε ένα τέτοιο σύστημα επιτήρησης και παρακολούθησης. Το κονδύλιο αυτό φυσικά δεν είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι μια καλή αρχή για την ε, εφαρμογή αυτού του συστήματος. Τέλος, συμφωνούμε με την εισηγήτρια σε ό,τι αφορά την διαθεσιμότητα των δεδομένων. Θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν, όπως κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι καλό παράδειγμα προς μίμηση οι Ηνωμένες Πολιτείες για την δωρεάν παροχή των δεδομένων που θα συγκεντρώσουμε από ένα τέτοιο σύστημα. Ευχαριστώ. Η Αμελή Αντερστότερ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που με βοήθησαν με τα σχόλιά τους και ευχαριστώ και την Επιτροπή για τους ίδιους λόγους. Θα ήθελα να πω ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα σας έχω δώσει ένα προσχέδιο της γνωμοδότησης και στις 14 Νοεμβρίου θα έχετε το τελικό σχέδιο. Στο μεταξύ θα έρθω σε επαφή με όλους τους σκιώδες και με την κυρία Καρβάλιο από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλό απόγευμα. Στις 14 Οκτωβρίου λοιπόν θα συζητηθεί ξανά αυτό το ζήτημα και η επόμενη συνεδρίασή μας προβλέπεται για τις 18 Σεπτεμβρίου ολόκληρη την ημέρα από τις 9 και από τις 3 μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία και σας χαιρετώ.